Συνάδελφοι, πριν αρχίσουμε, η κυρία Λίχτεμπεργκερ παρακάλεσε ε, στην ψηφοφορία να ψηφίσουμε πρώτα το θέμα των συμβάσεων γιατί πρέπει να φύγει, να πάει σε άλλη πολύ σημαντική επιτροπή. Ε, το σημείο 8 δηλαδή ε, είναι το πρώτο που θα ψηφίσουμε, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων αποφάσεις των συντονιστών, αν μου επιτρέπετε στα γρήγορα να σας τα πω. Άκουσαν τους εισηγητές ε, Κουμουτσάκου και Ερτούκ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών, για τις ε, τροπολογίες και συμφώνησαν οι συντονιστές ε, με τους εισηγητές να είναι λίγες οι τροπολογίες και να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια με ε, γνώμονα την ευρωπαϊκή προοπτική και προστιθέμενη αξία ορισμός εισηγητών. Συμφώνησαν οι συντονιστές να δώσουμε και νέους πόντους στις ομάδες ε, points στην επόμενη συνεδρίαση. Θα το συζητήσουν την επόμενη φορά οι συντονιστές. Σε ό,τι αφορά τώρα τις τρεις εκθέσεις σχέδιο ε, κανονισμού ε, για τους δρόμους για το ΕΛΚ, το δεύτερο ε, για τις επιθεωρήσεις επιτόπου και για τα εμπορικά αυτοκίνητα, όχι για γιοταχή σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι θα κάνουν την τρίτη έκθεση. Πρόταση οδηγίας που θα τροποποιεί την τρέχουσα οδηγία για την καταχώρηση και τα σχετικά έγγραφα ε, των αυτοκινήτων. Επίσης οι συντονιστές ε, σχετικά με την οδηγία 59 του 2003 για ε, τα επαγγελματικά προσόντα και την επαγγελματική κατάρτιση ε, δεν θα δοθεί η συνέχεια. Το ίδιο σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διοδίων και πάλι δεν θα κάνουμε τίποτα, ούτε συμφωνία με την Ελβετία για τα ευρωπαϊκά συστήματα πλοήγησης με δορυφόρων, ούτε για την πράσινη βίβλο ε, για τη χαρτογράφηση του βυθού των ωκεανών και σχέδιο ψηφίσματος από τον κύριο Ντεσιλβέστης ε, του ΕΛΚ σύμφωνα με τον, τον άρθρο 120 του κανονισμού. Δεν θα κάνουμε τίποτα επί του παρόντος, αλλά θεώρησαν οι συντονιστές ότι θα πρέπει το ψήφισμα αυτό να το εξετάσουμε στα πλαίσια της επόμενης έκθεσής μας για τις βιώσιμες αστικές συγκοινωνίες. Σε ό,τι αφορά το προγραμματισμό μας τώρα για το 2013, η απόφαση για τις αντιπροσωπείες έχει ε, ζητηθεί για τις Ηνωμένε Πολιτείε και Βορειοδυτική Αγγλία, Πολωνία και Πολογερμανικά σύνορα ε, είναι κάτι που προτείνουν το ΕΛΚ και οι πράσινοι και Σαρδινία είναι τα, τα άλλα δύο λοιπόν. Και αυτή ήταν η πρόταση των φιλελευθέρων. Για τις ακροάσεις, να σας δώσω και τις ημερομηνίες σας παρακαλώ για τις ακροάσεις. Σας δίνω τις ημερομηνίες να ξέρετε για να μην ακυρώνετε την προηγουμένη, όπως ήθιστε, οι Ηνωμένε Πολιτείε 11 Φεβρουαρίου, Βορειοδυτική Αγγλία, 29 Απριλίου και επόμενες ημέρες, Πολωνία, Πολογερμανικά σύνορα 15 Ιουλίου και Σαρδινία θα είναι η τελευταία αποστολή την Τυρκουάζ εβδομάδα της 28 Οκτωβρίου του 2013. Για τις ακροάσεις η απόφαση του Προεδρείου ήταν να πούν οι επιτροπές ποιες ακροάσεις θέλουν να κάνουν ένα χρόνο πριν. Ε, αυτό μας προβληματίζει και μας ενοχλεί και όλα στη, ε, στη διάσκεψη των Προέδρων. Ε, πάση περιπτώσει. Είναι τρελή αυτή η απόφαση. Πού να ξέρω ένα χρόνο πριν τι ακροάσεις θέλω να κάνω. Λοιπόν, αποφάσισαν οι συντονιστές να γίνουν έξι ακροάσεις. Αυτό δεν μας απαγορεύει να κάνουμε και άλλες σε περίπτωση που χρειαστεί. Ως εξή. Τέταρτο πακέτο για τους υδροδρόμους. Στην, σε ε, αερομεταφορές, επίσης ε, σε έκτακτες περιστάσεις. Θυμάστε τότε με το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Τι θα γίνει αν εκραγεί άλλο ηφαίστειο, ξέρω εγώ, πάλι στην Ισλανδία εφαρμογή της τρίτης οδηγίας για τις ε, ταχυδρομικές υπηρεσίες, λιμενικές υπηρεσίες, μέγα τράξ, αυτά τα μεγάλα φορτηγά και τέλος βελτίωση των ε, εσωτερικών πλωτών οδών και των διασυνδέσεων. Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας εγκρίθηκε και πρέπει να κυκλοφορεί αυτή την ώρα. Σημειώστε παρακαλώ ότι έχουμε μια-δυο πέμπτες, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, δεν μπορούμε να τις ε, καταργήσουμε όλες είναι η ποσόστοσή μας να έχουμε συνεδρίαση την πέμπτη ολόκληρη. Το μοιραζόμαστε αυτό με άλλες επιτροπές. Και θα ήθελα να σας πω ότι το απόγευμα πότε είναι, 9η Οκτωβρίου είναι. Ακυρώνεται. Πότε ήταν, ε, για πέμπτη απόγευμα. Της ε, Επιτροπής Μεταφορών τον Οκτώβριο. Α, όχι, τρίτη απόγευμα. Στην επόμενη συνεδρίασή μας έχει ακυρωθεί. Επιτροπολογία, newsletter, κυκλοφορεί και το προηγούμενο και στα διάφορα ακυρώθηκε, η Παμινάτη Οκτωβρίου το απόγευμα και η γραμματεία θα σας μοιράσει ε, ενημέρωση ε, για τη δυνατότητα να ζητήσουμε και νέες μελέτες από τον προπολογισμό του 2012. Έχουμε κάτι λεφτά που περισσεύουν και υπάρχει χώρος να γίνει μελέτη αν επιθυμούν κάτι τέτοιο και έχουν ιδέσει οι πολιτικές ομάδες για το τι θα μελετήσουμε. Ερωτήσεις έχετε για όλα αυτά που σας είπα. Θα σας δώσουμε και τα πρακτικά, ε, μάλλον όχι και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων για το 2013 το συντομότερο. Ευχαριστώ πολύ και περνούμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Ποιος δεν έχει κάρτα. Γιατί ε, δεν βρίσκει ο Αλχαντράου την κάρτα του, γιατί είναι μπλεγμένη μέσα σε κάτι πενιντάρικα εκεί πέρα. Τόσα λεφτά που έχει, πού να βρει κάρτα. <laughs> Mr. has not got his voting Λοιπόν, ο κύριος Αλχαντράουι δεν έχει κάρτα. Ο μοναδικός μέχρι στιγμής. Άλλον, έχουμε. Όχι. Hey, can we do a, check down the... Λοιπόν, να κάνουμε έναν έλεγχο. Αρχίζει ηλεκτρονική ψηφοφορία για να ελέγξουμε τις κάρτες. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εντάξει, δεν υπάρχει υπεράριθμος από καμία πολιτική ομάδα, είμαστε εντάξει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον κύριο Αλ Καντράου και τον κύριο Μπάνκι χωρίς κάρτα, αυτοί οι δύο. Ωραία. Να μας λέτε κάθε φορά, σηκώνοντα το χέρι, τον αντίχειρα, τι θα ψηφίσετε. Πρώτη, είπαμε, θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Λίχτεμπεργκε που ήταν το 11 Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων, είναι σχέδιο γνωμοδότησης για την πρόταση οδηγίας για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Η τροπολογία 1 της εισηγήτριας. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. δύο ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. 43 ζήλε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να το ελέγξουμε παρακαλώ. Την 45 ηλεκτρονική επαλήθευση που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 ψήφι κατά απόχες εγκρίνεται η 4 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η 5 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η 6 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ. Όχι, να πάμε στην 11 λέει. 11 υπέρ, οι άλλες έχουν καταπέσει. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά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 αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ τσεκ. Ωραία, ελέγχουμε τη 12 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Κύριε Μπάνκη, εσείς, κατά. 21 ε, υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. 66 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 20 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 68 είπε, κατά αποχές απορρίψεται. 69 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 22, 23, 24 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Να το ελέγξουμε παρακαλώ αυτό. Συμβιβαστική α. Ηλεκτρονική επαλήθευση. As όλοι ένας ε, υπέρ, ένας κατά, χωρίς κάρτα, πέρας. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 είναι συμβιβασμός με ψηφοφορία κατά τμήματα τα εξή τρία. Τμήμα πρώτον. Όλο το κείμενο χωρίς κόστος παραγωγής και ε, κοινωνικού αντικτύπου. Το δεύτερο είναι το κόστος παραγωγής και το τρίτο είναι το κόστος κοινωνικού αντικτύπου. Τα καταλάβατε? Ωραία. Ψηφίζουμε το πρώτο. Τι συμβιβασμό είναι αυτός με split vote, εν Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ το πρώτο τμήμα. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ένας υπέρ, ένας κατά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας απορρίπτεται με ισοψηφία. Άρα το σύνολο του συμβιβασμού απορρίπτεται. Οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε τα υπόλοιπα. Και πάμε τώρα στην 78. Όχι, συγγνώμη, 77. Το κύριο Ζήλε, ψήφιπε Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 77, αρχίζει η ψηφοφορία. το όλοι. Πέρας. Το αυτό. Με την ίδια ισοψηφία. Απορρίπτεται. 76. Ψήφι υπέρ. 76. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 επέ, κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεν ψηφίσουμε την 27 28 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 32. Για το άρθρο 62 παράγραφος 2. 69 συγγνώμη παράγραφος 2. Ψηφίσουμε 32 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα. Την 32 παρακαλώ. Στο άρθρο 69, 2. Ψηφίζουμε τροπολογία 32. Έχουμε ένα κατά και έναν υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. Πάμε στην 33. Υπέρ κατά, αποχές, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 33. Ψηφίζουμε τώρα. Συν μία ψήφος υπέρ και μία κατά. Πέρας προφορίας. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 89 ως προσθήκη υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 90. Ψηφοφορεί κατά τμήματα σε δύο τμήματα. Πρώτο, χωρίς το however μέχρι το the contract. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται επίσης. 35. Το υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 36. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 92. Υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 37. Τώρα ψηφίζουμε. Συν μία ψήφος υπέρ και μία κατά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39, 95 και 47 μαζί υπέρ κατά αποχές υιοθετούνται. 98. Α, όχι, ήταν και 98 μαζί με τις προηγούμενες, έτσι. 96 τώρα, υπέρ. Κατά. Απόχες, απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 και 67 μαζί, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτονται. 104 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Σα... Κατά, αποχές υιοθετείται. 41 υπέρ. Κατά, αποχές υιοθετείται. Και 42 υπέρ. Κατά, αποχές υιοθετείται. Και Τελική ψηφοφορία τώρα. Ξεκινάει η ψηφοφορία παρακαλώ. Συν δύο ψήφοι υπέρ με τον κύριο Μπάνκι. Ψήφισαν όλοι. Υιοθετείτε. 36 υπέρ. 4 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Λίχτεμπεργκερ. Μάλιστα. Μικρό διάλειμμα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Έρθω να βγάλω το φακελάκι με το τσάι που το είχα στην τσέπη, έτσι για να είμαι έτοιμο όταν έρθει το τσάι. Αν ε, αρχίσω να κραδένω το, το σακουλάκι θα σας τάσει και η μυρωδιά. Πάμε στην επόμενη έκθεση Λίχτεμπεργκερ. Sorry, Eva. Συγγνώμη, Εύα, τα έμπλεξα εδώ. Τροπολογία 2. Ε, το time, Mike. 2. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τη 2. Τώρα ψηφίζουμε. Νομίζω ότι περνάει, αλλά ας το ελέγξουμε. Ψήφισαν όλοι. Είστε σίγουροι. Ελάτε λοιπόν, ψηφίστε. Πέρα τη συν μία ψήφο υπέρ και μία κατά, υιοθετείτε. Τρία. Υπέρ. κατά. Αποχές υιοθετείτε. Πάμε στις 40 τώρα. Ε, Μάικλ, ξέρεις ότι για μας τους Βρετανούς το, το τσάι είναι προτεραιότητα. Πάμε στην uh, τροπολογία 40. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές, υιοθετείτε. Η 54 καταπίπτει. Όχι, όχι, όχι. Δεν καταπίπτει. Υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ. Ψηφίζουμε. Κατά τώρα. Αποχές. Να την τσεκάρουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Συν μία ψηφός υπέρ και μία κατά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Ξανά. Μπορούν να ψηφίσουν και οι σοσιαλιστές. Την τέσσερα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 42. Υπέρ. Θέλετε να τσακάρουμε τη 41. Ψηφίσουμε τώρα τη 41 ηλεκτρονικά. Συν 2 ψήφι υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Θα μπορούσαμε τα είχαμε κάνει μαζί όλα αυτά. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 13 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 50 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά αυτό το σημείο, την 50 δηλαδή, τροπολογία 50. Μία ψώση υπέρ και μία κατά. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 51 της Μάισνερ υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 52 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 52 ψηφίζεται μία ψήφος υπέρ, μία ψήφος κατά επιπλέον, πέρας ψηφοφορίας, υιοθετείται 53 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 14 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 15 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 16 υπέρ, κατά αποχές υιοθετείται 17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 19, 20 και 21 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 22 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Συμβαστική γάμα με ψηφορικά τμήματα σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 56. Ζήλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ υπέρ της 25 κατά Εποχές υιοθετείται 26 υπέρ Πάμε στην 29. Οι άλλες καταπίπτουν και η μία έχει αποσυρθεί. Άρθρο 79, παράγραφος 2, τροπολογία 29. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 32. Υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 33 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 35 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 61 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 36 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 36 υπέρ κατά Μόλις την ψηφίσαμε. Να μην την ξαναψηφίσουμε. 62 και 63 μαζί. 64-65 επίσης. Μαζί, έτσι. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 62, 63, 64 και 65. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τώρα. Μετράμε και μία ψήφο υπέρ, μία ψήφο κατά. Επιπλέον. Πέρας φοφορίας. Υιοθετούνται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένα, Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Και 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Και δύο ψήφοι υπέρ. Προστίθενται. Πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείτε 37 ψηφιπέρ κατά, 4 κατά. Μπράβο κυρία Λίχτεμπεργκ. Όχι, όχι, λάθος έκανα πριν. 38 ψηφίπερ υπέρ, 3 ψήφι κατά. Και τώρα πάμε στην έκθεση Μπαχ. Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα κουραστώ, γι' αυτό θα ήθελα να ψηφίσετε καλά και διάκριτα. Ξεκινάει μαραθώνιος. 15, που είναι γλωσσική αλλαγή για το γερμανικό κείμενο. Όχι, για το αγγλικό. το εδώ λέει γερμανικό. Να το ψηφίσουμε, δηλαδή. Όχι, όχι, γλωσσικό είναι αυτό το σημείο. Πάμε στα 16. Κόζα. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 21. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. Συμβασμός υπάρχουν δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. Περνάει και ένα συμβασμός επιτέλους. Γυρνάμε τη σελίδα. Πάμε στην ε, τροπολογία 28 Taylor. Υπέρ κατά αποχές τσεκάρουμε την 28 μια ψήφος υπέρ μια κατά επιπλέον ψήφισαν όλοι πέρας φοφορίας υιοθετείτε 29 Τέιλορ υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε 30 υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 35 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε 37 ηλεκτρονικά. Μια ψήφος μια... Δεν μετράμε άλλες ψήφους τώρα, για... μόνο μία μάλλον, γιατί ο άλλος έχει την κάρτα του ο άλλος βουλευτής. Είναι ισοψηφία, αλλά απορρίπτεται γι' αυτό. 38 του Δανέλη, υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται. 39, υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, εποχές υιοθετείται. Σαράντα, Ρικέ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 43. Για το πρώτο καλύπτεται το συμβασμό. Σαβισάρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 55. Έχει αποσυρθεί αυτή. 56 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 58 υπέρ κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 59 υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 60 υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 61 υπέρ, κατά, αποχές. Τσεκάρουμε την 61 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε τώρα. Συνία υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Υιοθετείτε. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 80. Υπέρ. Κατά αποχές υιοθετείται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 102 καταπίπτει γιατί 81 πέρασε. Πάμε στην 82. Κοχ, υπέρ, κατά, εποχέ υιοθετείται. 83 που είναι γλωσσική αλλαγή. Χρειαζόμαστε μία τροπολογία για να αλλάξουμε την αναφορά στη Γενική Διεύθυνση MOVE. Να το κάνουμε δηλαδή Γενική Διεύθυνση MOVE αντί για τρέν. Ψηφίζουμε την τροπολογία λοιπόν. Έτσι, υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε, 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 89 99, μάλλον 99 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 116 καταπίπτει αυτή 117 επίσης και 140 πίπτη και πάμε στα 100. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 102, Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείτε. 103 καταπίπτει αυτή. Το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Πω, πω, πω, πω, πόσο το περιπλέξατε το πράγμα. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 104. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 105 η επόμενη υπέρ, κατά, αποχές. Θα το ξαναπροσπαθήσουμε. 105 υπέρ, ευχαριστώ. Κατά, αποχές, υιοθετείτε. 106 και πάλι μια γλωσσική αλλαγή. Λοιπόν, ψηφίζουμε για το 106 υπέρ, Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 107. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Συνεχίζουμε να ψηφίζουμε για αυτήν. Ρωτάει ο πρόεδρος. Άρα έχουμε υιοθετήσει την 106 Είναι μια προστίκη λοιπόν για το 107 υπέρ. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές Υιοθετείτε. 112 και έχουμε και μια προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ε, αντιρρήσεις στην προφορική. Όχι, επομένω το συμπεριλαμβάνουμε υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 113 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121, 22 και 24 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Προχωράμε στην 125, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 126 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. υιοθετείται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, υιοθετείται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 131 εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά Αποχέ. υιοθετείτε. 143 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 144 και 145 είναι ίδιε υπέρ κατά Αποχέ. υιοθετούνται. 146 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτονται. 147 υπέρ Ελέγχουμε την 146, έναρξη ψηφοφορίας για την 146. Ψήφισαν όλοι, συν 1. Μία ψήφος υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. Και υιοθετείται. Καλά που ελέγξαμε. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 148. Καταπίπτει 149 επομένως υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, ε, υιοθετείται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 αυτό είναι ε, συμπληρωματική προς την ε, συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, Αποχές υιοθετείται. 156 και πάλι ε, υπάρχει και προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική. Ο κύριος Ναι, έχουμε μια αντίρρηση. Επομένω δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία. Άρα είναι η αρχική τροπολογία ως προσθήκη στην 7 συμβαστική υπέρ κατά αποχές, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ε, έναρξης ψηφοφορίας. Μία κατά συμπληρωματικά, πέρας ψηφοφορίας και υιοθετείται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείται. 159 της κυρίας Τικάου. Εκα... Υπέρ για την 159, κατά, αποχές, νο... Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, νομίζω ότι απορρίπτεται έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Συμβεβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 167, συμπληρωματική, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169, και πάλι, συμπληρωματική, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. Συμβιβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 176 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 172 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 177 λοιπόν και 178 μαζί είναι υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 180 κύριου Τέιλορ, υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 181. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 183. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Υιοθετείτε. 184. Σιαναλόβα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 186. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. συμβιβαστική 10, κατά, υιοθετείτε. 193 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 194 συμπληρωματική υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Υποθέτω ότι αυτό <laughs> σημαίνει ότι με παρακαλείτε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά και έναρξη ψηφοφορία. Συν ένα από τον κύριο Αλκατράουι. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Και απορρίπτεται. Θα έπρεπε να φωνάξω ζήτω τώρα, έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων 197 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 196 κατά αποχές υιοθετείται 22 δηλαδή ως συμβαστική 11 συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ...204 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 206. Με προφορική τροπολογία υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν όχι, μαζί με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται 207 και 209. Υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετούνται. 210, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Και τώρα συνεχίζουμε με το συμβασμό 12 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Και τώρα 2.17 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 2.18 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 2.20 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. 2.21 με ψηφοφορία κατά τμήματα. στο, το πρώτο μέρο καταπίπτει εξαιτία του συμβιβασμού 11, επομένω ψηφίζουμε για το δευτερο μέρο μέρος υπέρ. αποχέ, αποχές, υιοθετείτε. 2-2-3 υπέρ, κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. 2-24 υπέρ, κατά, αποχέ, υιοθετείτε. 2-25 υπέρ, κατά, Αποχέ. υιοθετείτε. 2-26 υπέρ, κατά, αποχές, Υιοθετείτε. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 229 είναι συμπληρωματική υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 2.32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και τώρα ε, στο 4. Citations. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τώρα συνεχίζουμε με τον 3. Κυρία Σάβησα. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Υιοθετείτε. Πέντε και έξι. Τα τρία, πέντε και έξι είναι τα ίδια. Επομένως έχουμε ήδη ψηφίσει. Εφτά από τον κύριο Κόζα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Συμβιβασμό 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ελεκτρονικό έλεγχο για το 12. Έναρξη ψηφοφορία. Ένα κατά από τον κύριο Αλκατάβη. Έχουν ψηφίσει όλοι πέρα ψηφοφορία Και υιοθετείτε. 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Με την ίδια πλειοψηφία υιοθετείτε 14. Κατά. Αποχέ. υιοθετείτε. Και τώρα συνεχίζουμε με τι τροπολογίε από την ΙΜΚΟ. Παραγραφό 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ. υιοθετείτε. Παραγραφό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονικό έλεγχο για την παράγραφο 2, έναρξη ψηφοφορία. ένα υπέρ. Συν. Ψήφισαν όλοι, πέρα ψηφοφορία Και απορρίπτεται. Παράγραφο 3 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Παράγραφο 4 Το μόνο που μπορούμε να ψηφίσουμε είναι η τελευταία πρόταση γιατί το υπόλοιπο καλύπτεται από τον Συμβασμό 2 για την τελευταία πρόταση υπέρ κατά υιοθετείται. 6, παράγραφος 6, υπέρ, κατά, αποχές υιοθετείται, 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 11, υπέρ, Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται και ποιο θα είναι το επόμενο 26 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές υιοθετείται 30 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται ο κύριος Μπακ πριν την τελευταία ε, τελική ψηφοφορία. Ja, ich stelle mir die Frage... τώρα το εξή. Έχουμε με ψηφίσει τροπολογίες γλωσσικές. Ε, γιατί δεν ψηφίσαμε την πρώτη του Ντίτερ Χόγκοχ την υπαριθμό 15, αφού άλλες γλωσσικές τις ψηφίσαμε. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να ξαναγυρίσουμε, γιατί είχαμε μπερδευτεί λιγάκι με τις γλωσσικές αλλαγέ και για το κατά πόσον ήταν μια γλωσσική αλλαγή και μόνο ή όχι. Είναι η οχι ειναι η στην πρώτη σελίδα είναι η 15, τροπολογία 15. Είχαμε συζητήσει κατά πόσον είναι ε, γλωσσική και μόνο ή όχι. τέλο πάντων, ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχέ. Υιοθετείτε. Ωραία λοιπόν. Το λύσαμε αυτό. Τελική ψηφοφορία, έναξη ψηφοφορία. Ο κύριο Αλκατράουι ψηφίζει υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Και Υιοθετείται με 43 υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Μπακ. Περνάμε τώρα στο MFS το στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς να αλλάξουμε βάρδια στο Προεδρείο, ρωτάει. Just recharge your arms for the MFF vote. Ετοιμαστείτε να σηκώνετε και πάλι ψηλά τα χέρια σας σε αυτήν την ψηφοφορία. Okay. Amendment 2, Mrs. Ayala. Τροπολογία 2, υπέρ κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 3, συμπληρωματική υπέρ, κατά, Αποχέ. υιοθετείται. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, Αποχέ. υιοθετείται. 5, Durant, υπέρ, κατά, αποχε απορρίπτεται. 6, Τικάο, υπέρ, κατά, Αποχέ. υιοθετείται. 7, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 8 υπέρ. Κατά. αποχή Υιοθετείται. 9 υπέρ. Κατά. αποχέ. Ελεκτρονικό έλεγχο για την 9. Έναρξη ψηφοφορία. Κατά ο κύριος Αρκαντράου. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία και εγκρίνεται. Τροπολογία 10 καταπίπτει, η 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 ε, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Και συνεχίζουμε με τη 15. Υπέρ. Κατά. Απο... Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15. Ένα της ψηφοφορίας. Κατά. Ο κύριος Αλκαντράουι και ε, πέρας ψηφοφορίας. Υιοθετείται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές υιοθετείται. 17 συμπληρωματική υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 18 με την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ε, με την προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 19 συμπληρωματική υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 21 ψηφοφορία κατά τμήματα. Για το πρώτο μέρος, ε, η φράση τα shall και τα λοιπά μέχρι National Allocations, για το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείται. Η 20 είχε αποσυρθεί. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 24. Κύριε Τουάν. Υπέρ. Κατά. Ε, ε, απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 28. Υπέρ κατά, αποχές, υιοθετείτε. 29 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 30 υπέρ, κατά, αποχές, υιοθετείτε. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα, αλλά έχει αποσυρθεί το πρώτο μέρος, επομένως δεν υπάρχει πρώτο μέρος και δεν είναι και κατά τμήματα η ψηφοφορία που θα κάνουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα και το μόνο που έμεινε υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 34 υπέρ κατά αποχές υιοθετείτε. 37 κατά πίπτη 35 υπέρ κατά ε, υιοθετείτε. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Και τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Υιοθετείτε. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη ψηφοφορίας. Και συνένα. Από τον κύριο Αλκαντράουι. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Και υιοθετείται, εγκρίνεται με 36 υπέρ, μία κατά και 5 αποχές. Η επόμενη... Είναι η έκθεση κυρίας Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλάξαμε βάρδια. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι καταπληκτούν οι δύο επόμενες. Πάμε στη 33 Κατά. Αποχές. Μπορούμε να αλλάξουμε παρακαλώ τη 33 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Για ψηφίσατε όλοι. Ένας υπέρ, ένας κατά επιπλέον. Πέρας. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 αρχίζει η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 35. Ψήφισατε όλοι. Συν μία του Σαΐτ Αλχαντράουι, πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Όχι, δεν είναι ισοψηφία γιατί είπαμε συν μία ψήφο του κυρίου Αλχαντράου που δεν έχει κάρτα. 36 ε, επόμενη υπέρ κατά άποχες έλεγχος για την 36. Βλέπω ότι κουράζεστε τα χέρια σας, ε, δεν τα σηκώνετε. Συν μία ψήφο, έτσι, ψηφίζουμε την 36 υπέρ Συγγνώμη, ηλεκτρονικά, πέρασε. Απορρίπτεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Η ε, επαλήθευση. 38. Της κυρίας Ντυρά. Αρχής ψηφοφορία. Συν μία. Ψήφος υπέρ Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 39 της κυρίας Ντυρό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος γιατί 39. Αρχίζει τώρα. Και πάλι σημεία του κυρίου Αλχαντράουι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία. 40 υπέρ. Μια στιγμή οι σοσιαλιστές και δημοκράτες ε, ψηφίστε και εσείς τη 40 υπέρ, κατά, άποχες και πάλι έλεγχος χρειάζεται νομίζω με την ίδια πλειοψηφία αλλά επειδή είναι πολύ σφιχτή ε, ψηφίζουμε τις 40 είναι ένα υπέρ τον κύριο Αλχαντράουι να ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 41. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 του εισηγητή περ, συγγνώμη της εισηγήτρας κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 Πε. κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην 56 προσθήκη στη συμβαστική 2 χωριστή σε τμήματα, δύο τμήματα. Το πρώτο είναι όλο το κείμενο χωρίς τον αέρα, σε άπνια δηλαδή, και η δεύτερη είναι με τον αέρα. 56 λοιπόν χωρίς τον αέρα είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα Α, τώρα ψηφίζουμε τον αέρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν μας αρέσει ο αέρας, σε πάση Ναι, αδικία λέει κάποιος. Ε, η προφορική ένα της κυρίας Αγιάλα ε, ως προσθήκη καταρχήν διαφωνεί κανείς με την προφορική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ως προσθήκη συμβαστική 2 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 62 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ο κύριος Αλκαντράου είναι κατά ψηφίσατε όλοι πέρασε Εγκρίνεται. 63 της κυρίας Ντουρό Ειπέ. κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στην 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την 72 λοιπόν αρχίζει η ηλεκτρονική υπολήθευση ο κύριος ε, Χαντράου είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 74. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 75. Αρχίζει η ψηφοφορία. Συν μία ψήφος υπέρ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 76 της κυρίας Ντουιρό. Ψηφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 τι εισηγήτριας υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική 4 ψήφι υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Επόμενη είναι 85. Υπέρ. Όχι, μια στιγμή. Ναι, ναι, 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. πίπτη. Συγγνώμη. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται ή 87. Όχι, 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 καταπίπτει. Η 14 της εισηγήτριας ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 91 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε αυτό. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Αρχίζει λοιπόν για την 91. Ο Σέντιν είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 92 σε ένα λοβά υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. «93 κατά τμήματα» μέχρι τους δείκτες επιδόσεων. το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η προφορική 2 της κυρίας Αγιάλα διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία όχι δεν ψηφίζουμε τότε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ καταπέφτει. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται 102 είπε, κατά αποχές να την ελέγξουμε παρακαλώ την 102 νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά η μικρή διαφορά συν μία ψήφος του κυρίου Ελχαντράου υπέρ ψηφίσατε πέρασε εγκρίνεται 21-20 18 της εισηγήτριας ψηφιπέ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές να την ελέγξουμε από αυτή παρακαλώ. 103. Αρχίζει ηλεκτρονική επαλήθευση συν μία ψήφος υπέρ του κύριου Αλχαντράουε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Αυτή η ψηφία Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία αρχίζει ηλεκτρονικά μία του κυρίου Ελχαντράουη και ψηφίσατε όλοι κλείνει 39 υπέρ, 4 κατά μία αποχή εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γκρισμπέκ. Στο επόμενο σημείο. Βοηθήστε με λιγάκι με το δεύτερο σημείο που είναι υπηρεσία εδάφου στα αεροδρόμια της Ένωσης και κατάρριση της οδηγίας ε, είναι η έκθεση Ζασάντα. Ο κ. Ζασάντα θέλει να κάνει μια παρουσίαση PowerPoint. Ε, δεν συνηθίζεται. Τώρα δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Όταν οι εισηγητέ παρουσιάζουν τι εκθέσει του, δεν συνηθίζουμε να κάνουμε τέτοιο τύπου παρουσιάζει. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Uh, δεν θα πάρει παραπάνω από το σύνηθες. Απλώς για να περάσει το μήνυμα, έτσι, και να, να είναι πιο σχηματικό, πιο απλό. What I'll do on this... Ωραία. Θα επιτρέψω την παρουσίαση PowerPoint να υπενθυμίσω στους βουλευτές όμως ότι δεν συνηθίζεται οι εισηγητές να κάνουν τέτοιες παρουσιάσεις στην Επιτροπή. Αυτό γίνεται σε ακροάσεις, σε άλλους χώρους, σε άλλα βήματα. Εδώ θα το επιτρέψω, αλλά κάνω έκκληση στους εισηγητές ότι άλλη φορά δεν θα μ' αρέσει, δεν θα είμαι έτσι τόσο χαλαρός και δεν θα επιτρέπω τέτοιες παρουσιάσεις PowerPoint. Κύριε Ζασάντα. Ξεκινήσετε, θέλ... θέλει να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι υπηρεσίε εδάφου στα αεροδρόμια της Ένωσης Αυτό είναι ένα σημαντικό κείμενο. Πού πήγαν οι διαφανειές μου, πού πήγε η παρουσίασή μου. Ας συνεχίσω. Αφορά χιλιάδες ευρωπαϊκά αεροδρόμια και πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας στα αεροδρόμια αυτά. Ετοιμάζοντας το έγγραφο εργασίας, Ήθελα να το παρουσιάσω και απλό αλλά και πλήρες για τους μελλοντικούς χρήστες. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το κείμενο, παρατήρησα ότι συχνά η συζήτηση το στο να συζητάμε θέματα απλώς απελευθέρωσης. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο του κανονισμού, αλλά δεν είναι το μόνο. Ε, ένα άλλο στοιχείο είναι η η ομοιομορφία των διαδικασιών και τα ελάχιστα πρότυπα στα αεροδρόμια. Διερωτώ μου λοιπόν πώς θα μπορούσα να δείξω με απλό και εύληπτο τρόπο με τι μοιάζουν διαδικασίες ε, που αφορούν τις υπηρεσίες εδάφους αεροδρόμια. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω γι' αυτό, για αυτές τις διαδικασίες. Πώς θα, με τι θα μοιάζει η εταιρεία, καταρχάς, που θέλει να δώσει τέτοιες υπηρεσίες. Ένας επιχειρηματίας που θέλει να κάνει τέτοιες υπηρεσίες, να δώσει τέτοιες υπηρεσίες σε δάφους αεροδρόμια, θα πρέπει να πάει στο κράτος μέλος και να πάει στο κατάλληλο φορέα για να εγκριθεί. Η διαδικασία έγκρισης ε, εξηγείται πολύ λεπτομερώς στον κανονισμό. Αυτός, αυτή η αρχή του κράτους μέλους θα διαπιστώσει αν αυτή η εταιρεία που είναι καταχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, έχει την κατάλληλη πολιτική και τα κριτήρια ε, για την ε, κατάρτιση του προσωπικού. Θέλω να απλουστεύσω τα πράγματα και θέλω να σας πω ότι κάθε ένας από τους φορέας στα κράτη-μέλη θα πρέπει να λειτουργεί με τον απλούστερο τρόπο, ούτω ώστε ο επιχειρηματίας να μπορεί να εγκρίνεται σε οποιοδήποτε ε, κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ισχύει μετά αυτή η έγκριση και στα 27. Ο επιχειρηματίας που παίρνει μια τέτοια άδεια ή έγκριση θα μπορεί να επιλέγει μετά το αεροδρόμιο που θέλει να προσφέρει αυτές οι υπηρεσίες από όλα τα αεροδρόμια που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή η έγκριση θα ισχύει για όλα τα αεροδρόμια. Θα είναι ενιαία, ομοιόμορφη. Σήμερα η διαδικασία έγκρισης είναι τελώ διαφορετική στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Έχουμε 27 διαφορετικέ διαδικασίε έγκρισης. Ο επιχειρηματίας θα πηγαίνει λοιπόν στα αεροδρόμια μετά για να μάθει ποια είναι τα ελάχιστα πρότυπα με τα οποία, τα οποία υπάρχουν και δεσμεύεται από αυτά. Τα ελάχιστα πρότυπα Υπάρχουν λοιπόν, και εδώ παρουσίασα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να τα παρουσιάσει αυτά τα πρότυπα με κατεξουσιοδότηση πράξης. Εγώ θα έλεγα ότι τα επιμέρους αεροδρόμια θα πρέπει να, έχουν, να αποφασίσουν, γιατί γνωρίζουν καλύτερα και εδώ πέρα υπάρχουν καμιά δεκαριά περιπτώσεις, ε, κατηγορίες ας πούμε, που τις βρίσκεται σε παράρτημα στον κανονισμό. Εδώ αυτές περιγράφουν, κάθε κατηγορία δηλαδή περιγράφει με, κάποια, με κάθε λεπτομέρεια το αεροδρόμιο και λέει, ας πούμε, τον ελάχιστο χρόνο για, την, για το check-in των ε, βαλιτσών για την πρώτη βαλίτσα, για την τελευταία βαλίτσα, για το πώς ελέγχεται τη βαλίτσα. Και πολλές άλλες κατηγορίες που βλέπετε εδώ. Μερικά από αυτά που αναφέρονται εδώ, νομίζω ότι θα κάνουν μερικούς να χαμογελάσουν, γιατί θα τους αρέσουν. Επίσης, τι επηρεάζει το περιβάλλον. Αυτά είναι κάποια από τα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να εισάγει το αεροδρόμιο, ούτω ώστε να αποκλειστεί περίπτωση απουσία ελέγχων. Επίσης, αυτά τα πρότυπα θα πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, το οποίο θα, που θα ελέγχουν, αν τα πρότυπα αυτά είναι πολύ ψηλά, πολύ αυστηρά δηλαδή, πολύ χαλάρα. όταν ένας επιχειρηματίας ξέρει ότι μπορεί να πληρεί αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, μπορεί να ψάξει, ε, μια, να βρει μια εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, ε, και αν η αεροπορική εταιρεία, ενδιαφερθεί για τις υπηρεσίες του, μπορεί να ξεκινήσει την επιχείρησή του. Ε, υπογράφεται η συμφωνία και εν συνεχεία ο επιχειρηματίας αρχίζει τη δουλειά του με βάση τα ελάχιστα πρότυπα και τη σύμβαση που υπέγραψε. Ο κανονισμός επίσης μιλάει για την ευκαιρία που υπάρχει να εξαιρεθούν σε ορισμένες χώρες κάποιες διατάξεις για την, που αναφέρουν την πλήρη απελευθέρωση. Σε ένα συγκεκριμένο τερματικό, ας πούμε, σταθμό, βλέπετε 11 κατηγορίες που αναφέρονται για δραστηριότητες υπηρεσιών ε, δάφους αλλά οι περιορισμοί μπορούν να αφορούν μόνο τέσσερι. Όλε οι άλλε κατηγορίε έχουν απελευθερωθεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορείτε να βάζετε περιορισμούς, δηλαδή στον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών. Αλλά για τις τέσσερις αυτές που βλέπετε με κόκκινο, ας πούμε για την παροχή καυσίμων, κυροζήνης και τα λοιπά, για το χειρισμό των αποσκευών και τα λοιπά, εκεί μπορεί λόγω του μεγέθους του αεροδρομίου να εισαχθούν περιορισμοί. Ε, τα αεροδρόμια με 2 με 5 εκατομμύρια ε, επιβατών μπορούν να έχουν δύο τέτοιους παρόχους υπηρεσιών. Αν έχετε 5 με 35 εκατομμύρια επιβάτες σε ένα αεροδρόμιο, Δεν μιλάω για τους τόνους εδώ, έτσι τα λέω πολύ απλά. Μέχρι τρεις παρόχους υπηρεσιών και τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη, για τα 7 μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη, μπορούμε να βάλουμε τον περιορισμό των τεσσάρων παρόχων υπηρεσιών κατά ελάχιστο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκάζεται οποιοδήποτε να πάει να δώσει υπηρεσία στην αεροδρόμιο. Εάν υπάρχουν δύο ε, πάροχοι και δεν υπάρχει τρίτος ή τέταρτος που να ενδιαφέρεται, κανένας δεν, πρέπει να τους, δεν μπορεί να τους αναγκάσει να ξεκινήσουν την παροχή υπηρεσιών εκεί. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν υπάρχουν 7 ή 10 που ενδιαφέρονται σε ένα κράτος μέλος να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, αλλά το κράτος μέλος λέει ότι αυτό το αεροδρόμιο, λόγω της υποδομής του, πρέπει να περιορίσει τον αριθμό των εταιριών παροχής υπηρεσιών εδάφους σε δύο, τρεις ή τέσσερις εταιρείες. Και τότε η διαδικασία προσδιορίζεται στο έγγραφο λεπτομερώς και όλη τη διαδικασία υποβολής προσφορών που θα επιτρέψουν την επιλογή των καλύτερων που μπορούν να δουλέψουν σε αυτό το δεδομένο αεροδρόμιο. Ήδη οι συνάδελφοι μου έκαναν διάφορες προτάσεις και γι' αυτό έχω βάλει στο έγγραφό μου μία διάταξη που λέει ότι ένα κράτο μπορεί να υποφεληθεί να, από την αναστολή της πλήρους απελευθέρωσης στα μεγάλα αεροδρόμια πάνω από 35 εκατομμύρια επιβατών δηλαδή μπορεί να αναστολεί το άρθρο αυτό για πέντε χρόνια που σε συνδυασμό με όλες τις άλλες δυνατότητες αναστολής ή εξαίρεσης για τερματικούς σταθμούς ή αεροδρόμια ολόκληρα, καθιστά κάποιες διατάξεις του κανονισμού ενισχύει, ενισχύει μόνο μετά από 10 χρόνια δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει, δεν πρέπει να εφαρμοστούν καθόλου, όχι βέβαια. Ξέρουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα, θα ισχύσει για τουλάχιστον 10 χρόνια. Όχι για 2, 3 ή 4 χρόνια. Για τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν. Θα ισχύει για μια μεγάλη χρονική περίοδο. Θα τελειώσω, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω περαιτέρω. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ε, ακούστηκαν απόψει ότι τέσσερις πάροχοι υπηρεσιών εδάφους σε αεροδρόμια είναι πολλοί. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας τα 7 μεγαλύτερα δρόμια ε, που καλύπτονται από αυτή τη διάταξη, δύο από αυτά έχουν πλήρη απελευθέρωση, τρία ακόμα είναι σχεδόν σε φάση πλήρους απελευθέρωσης και το πρόβλημα αφορά μόνο ακόμα δύο. Τα δύο που παραμένουν. Αναφέρεσουμε τα πέντε από τα εφτά. Αυτά τα δύο αδροδρόμια με τις διατάξεις του κανονισμού με τις διατάξεις για τους τέσσερις παρόχους υπηρεσιών μπορούν να αναστείλουν αυτή τη διάταξη για 10 χρόνια. Ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια και τις υποδείξεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέρνερ από την Επιτροπή Περιφερειών τώρα. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε κύριε Σίμψον. Κύριε σας... Μια στιγμή κύριε Βέρνερ. Τρία με τέσσερα λεπτά το πολύ έχετε. Αξιότιμο κύριε ε, Σίμψον, κύριε Σασάντο, ευχαριστώ πολύ ε, για το γεγονός ότι μας δίνετε την ευκαιρία να γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Περιφερειών και προφορικά εδώ. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε ούτε την υπομονή σας ούτε το χρόνο να καταχραστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ένα πακέτο για τα αεροδρόμια με τρία σχέδια κανονισμού και τα τρία αυτά τα είδαμε μαζί. Ε, και επίκειται και άλλη συζήτηση για τις χρονοθυρίδες, τα σλότ ε, που ε, έχουν μεγαλύτερη πίεση και οι αεροπορικές εταιρείες, ενώ αυτό που συζητούμε σήμερα αφορά μεγαλύτερη πίεση για τους αερολιμένες. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά ισορροπημένη η πρόταση η Επιτροπή Περιφερειών βλέπει θετικά στοιχεία για απελευθέρωση περαιτέρω της αγοράς και σε εμά στη λειψία στη Σαξονία που έχουμε μεγάλο αεροδρόμιο το βλέπουμε πώς αναζωογονείται και αναπτύσσεται η οικονομία. Ε, ε, μας ενώνει αυτός ο στόχος. Λέμε ναι λοιπόν ε, στην απελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφους, είναι θετικό, ενισχύει και την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα ε, γενικότερα. Λέμε όμως και κάτι άλλο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, οι δυνατότητες χωρητικότητας, προβλήματα χώρου, ασφαλείας. Αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Όπως είπε και ο κύριος Σαζάντα, να υπάρξει κάποια μεταβατική ρύθμιση για την τάξη μεγέθους ε, και του αεροδρομίου. Βέβαια, ε, αυτό δεν το προσδιορίζω ε, μπορεί να αφορά και μικρότερα αεροδρόμια, αλλά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες. Ο δρόμος προς την απελευθέρωση και το βήμα είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Μεγάλη πρόκληση. Έχουμε άλλα δύο σημεία που κάνουμε παρατηρήσεις. Το ένα είναι ότι θα πρέπει όλοι οι πάροχοι να μπορούν να κάνουν ε, και ε, συμβάσεις με ε, άλλες εταιρείες, ε, με υπεργολαβίες, όπως το λέει το άρθρο 35, και επίσης θα πρέπει τα αεροδρόμια να έχουν τη δυνατότητα επιβολής των κανόνων. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ο κανονισμός να είναι τόσο λεπτομερής, δεν είμαστε βέβαιοι. Συνοψίζω. Είναι καλό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ και πάλι που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε εδώ και προφορικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέρνερ. Οι πολιτικές ομάδες. Τέσσερα λεπτά συν τρία για τους υπολείπους. Ο κύριος Φλέκενστάιν από τους σοσιαλιστές και οι δημοκράτες Τέσσερα λεπτά και παρακαλώ να τα τηρήσετε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα όσα μας ε, παρουσίασε. σε μια πρώτη συζήτηση αξιολογήσαμε τα πράγματα, έχουμε κάποιες παρατηρήσεις. Για να αρχίσω από τα αρνητικά. Πρώτον, σε αντίθεση με εσά, κύριε Σεγητά και με τον προσκεκλημένο μας από την περιφέρεια της Λειψίας, εμείς δεν θέλουμε υποχρεωτικό επιπλέον αριθμό παρόχων. Θεωρούμε ότι με τους δύο τουλάχιστον παρόχους, όπως λέει η παλιά οδηγία, είμαστε εντάξει. Κάθε αεροδρόμιο μπορεί να απελευθερώσει τις υπηρεσίες ε, όπως θεωρεί σωστό και ε, πλεονέκτημα. Αλλά δεν, δεν ε, μπορεί κανείς να αναγκάσει κάποιον να είναι ευτυχισμένος από ένα ελάχιστο αριθμό παρόχων και μετά. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα του νομικού διαχωρισμού συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει νομικός ε, διαχωρισμός, αλλά λειτουργικός διαχωρισμός. Τι σημαίνει αυτό. Ε, χωριστή τήρηση βιβλίων. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν ε, ε, πλάγιες επιδοτήσεις του αερολιμένα προς τον πάροχο υπηρεσιών. Ξέρουμε τη συζήτηση που είχε γίνει για το unbundling, για την αποδέσμευση. Ε, πάντως η κατεύθυνση είναι σωστή. Σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, συμφωνούμε απολύτως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν, έχει, ε, δεν θα πρέπει να έχει εξουσία για της πράξης στο παράρτημά σας αναφέρεται ε, μια σειρά προτύπων, ε, θα τα ξανακοιτάξουμε προσεκτικά, αλλά θα δούμε και πώς θα πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση. Ε, και πάλι και εκεί μπορούμε κάπου να τα βρούμε για να συμφωνήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκρισης, μιλάτε για τις συλλογικές συμβάσεις. Εμείς θα θέλαμε και μια αντιπροσωπευτική ε, συλλογική σύμβαση. Εσείς μιλάτε για τις ισχύουσες συμβάσεις. Υπάρχουν κάποιες μικρές αποχρώσεις ε, σε αυτά τα θέματα, αλλά θα χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπεργολαβίες, εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει ε, οι πάροχοι του ίδιου του αερολιμένα να κάνουν υπεργολαβίες, ανάθεση σε τρίτους. Εκτός ε, βεβαίω ε, αν συμμετέχουν στο διαγωνισμό που είναι δημόσιος όπως και άλλοι. Όταν παραβιάζονται οι ελάχιστοι κανόνες ποιότητας θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία προσφυγής, θα πρέπει να το σκεφτούμε. Νομίζω ε, η πρώτη προσφυγή θα πρέπει να είναι η Επιτροπή Χριστών και η δεύτερη δυνατότητα προσφυγή στο κράτος μέλους. Εσείς προτείνετε πλήρη απελευθέρωση ε, της ίδιας ε, παροχής υπηρεσιών εδάφους, από το ίδιο το αεροδρόμιο δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί σε δύο ε, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ένα σημείο που δεν βρήκα στην έκθεσή σας, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε πώς πρέπει να το χειριστούμε αυτό, είναι το θέμα των δικτών. Πρέπει να πούμε και ε, γι' αυτό κάτι στην έκθεση αυτή, να το ξανασκεφτούμε και να το αποφασίσουμε. Δηλαδή, σε πολλά σημεία μπορεί να είμαστε στον ίδιο δρόμο, μπορούμε να συγκλίνουμε και να βρούμε συμβιβασμούς, Τώρα για το αριθμό των παρόχων 3 και 4 δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλίντς από τους φιλελευθέρους. Ε, τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα επιθυμούσα κανονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει προτεραιότητες και να ασχολείται με θέματα ε, όπως πώς μπορούμε να έχουμε ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, ένα αέριο χώρο και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν οι αεροπορικές μας εταιρείες. Βλέπουμε μια μετά την άλλη εμφανίζουν ελλείμματα. Οι αερολιμένες μια χαρά λειτουργούν. Το πρόβλημα είναι στις αεροπορικές εταιρείες. Η Qantas ε, ε, μόλις ε, ε, τα χάλασε με την British Airways και τα έφτιαξε με την Emirates. Λοιπόν, δεν ακούω να λέτε τίποτα για τις αεροπορικές μας εταιρείες. Επίσης θα ήθελα μια πρόταση για τους αερολιμένες ε, στην Ευρώπη ε, να ιδιωτικοποιηθούν όλοι, γιατί είναι κρατικοί σήμερα ή μη κρατικοί οι περισσότεροι. Αν γίνουν ιδιωτικοί, από μόνοι τους θα προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα τέτοιο μοντέλο επιχειρηματικό, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί. Οπότε δεν χρειάζεται εμείς να συζητάμε για τις υπηρεσίες εδάφους. Εμένα εξακολουθεί να με ενοχλεί το γεγονός ότι αυτό το θέμα το χωρίσαμε όπως χωρίστηκε και το μοιραζόμαστε δηλαδή στην Επιτροπή, εδώ τη δικιά μας με την Επιτροπή Απασχόλησης γιατί ε, πολλά από αυτά που κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις δικές μας εργασίες και όταν Ακούω τις προτάσεις εκεί στην Επιτροπή Απασχόλησης που θα τις ψηφίσουν ε, με πιάνει κρύωση κρύος υδρότας, διότι από τη μια υποτίθεται ότι είναι υπέρ της ε, απελευθέρωσης, αλλά θέλουν να περιορίσουν μαζικά ε, την ελευθερία του επιχειρήν. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν τα ανέχω. Συμφωνώ ε, σε πολλά με τον εισηγητή. Εγώ φιλελεύθερο είμαι, θέλω απελευθέρωση. Βεβαίω ελάχιστε προδιαγραφέ, αλλά μην τα ορίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι ίδιοι φορεί επιτόπου. Αλλά και εδώ έρχομαι σε αυτό που είπε προλαλή σας, γιατί πρέπει να είμαστε εμείς τόσο απόλυτοι. Εγώ ξέρω ε, το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης γιατί μένω εκεί κοντά δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνει κανείς τίποτα. Ακόμα και με ε, τον τρίτο διάδρομο προσγείωσης είναι δύο οι ε, πάροχοι υπηρεσιών και ε, μπουρδουκλώνονται μεταξύ τους. Ε, ε προ, έρχονται διάφορα λεωφορεία δεξιά και αριστερά ε, που είναι δύο. Φανταστείτε να υπήρχε και τρίτος και τέταρτος. Χαιρετίσματα. Ε, αυτό βελτιώνει την ποιότητα για τον καταναλωτή ή τον επιβάτη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επί της αρχής, ναι, στην ενιαία διαδικασία Ακόμα και κάποιος είναι εγκεκριμένο ως πάροχος σε μια χώρα, θα πρέπει αυτόματα να μπορεί να λειτουργεί και σε άλλη χώρα της Ένωσης. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση εκεί που κάνουν την ίδια την υπηρεσία, τα αεροδρόμια τα ίδια, θα πρέπει να χωριστεί αυτό. Δεν ξέρω όχι μόνο λειτουργικά αλλά και νομικά. Βεβαίως να είναι απόλυτο ταμπού και να απαγορεύονται οι πλάγιες επιδοτήσεις, οι υπόγειες ε, και για την ε, κατάρτιση, μετεκπαίδευση και αυτό είναι αυτονόητο. Εμείς πρέπει να το πούμε αυτό νομοθετικά. Αυτό είναι ουσιαστικό τμήμα της παροχής υπηρεσιών. Και αυτοί οι πάροχοι ήδη γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να είναι πραγματικά ε, στην αιχμή ε, του δόρατος. Τώρα για τους διαγωνισμούς και ε, η διάρκεια των συμβάσεων είναι επταετής, δεκαετής. Καλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, ούτε το αποφασιστικό. Σφυράκι τέλειωσα. Εντάξει. Πάντως θα συμφωνήσουμε νομίζω κύριε Σασάντα. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο σκιώτης μας ηγητής είναι ο Πίτερ Βαντέλα. Δυστυχώς δεν μπορέσει να έρθει, γιατί ε, οργανώνει την ε, Ολλανδική κυβέρνηση, μάλλον. Ευχαριστώ όμως τον εισηγητή για όλη την προσπάθεια και μου έδωσε να πω δύο-τρία σημεία. Κάποια από αυτά τα είπαν οι συνάδελφοι για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητα. Έχουν ήδη οριστεί. Θεωρούμε ως ομάδα ότι υπάρχει επίσης ένα θέρμα αμοιβαία αναγνώρισης και ανταγωνισμού με τρίτες χώρες. Κυρία Ζασάντα, θα σας δώσω ένα κατάλογο με τα θέματα που θέλει να θέσει. Επίσης, οι νέες κατηγορίες αεροδρομίων, δεν συμφωνούμε με αυτές. Τρία, τέσσερα σημεία, πέντε τέλο πάντων. Εμείς όμως στην ECR εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα και το Μάρτιο η συνάντηση του Συμβουλίου ε, υποστήριξε τη γενική προσέγγιση πάντως. Και εμείς την υποστηρίζουμε και στον Ομένο Βασίλειο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε κάποια στοιχεία του προτινόμενου κανονισμού. Εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει απελευθέρωση, δούλεψε καλά. Αν κοιτάξετε κάποια αεροδρόμια, έχουν διάφορους, αρκετούς παρόχους υπηρεσιών και λειτουργήσε καλά το πράγμα. Δεν θέλω να παροθέσει, αλλά το θέμα της Φραγκούρτης είναι ένα ζήτημα βέβαια και θα πρέπει να επιληθεί. Αλλά τελικά η συζήτηση γυρνάει γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος. Ε, μπορεί να υπάρχουν μικρότερα αεροδρόμια που μπορεί να μην είναι απελευθερωμένα, που μπορεί να είναι στα χέρια των αρχών. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρούμε την ισορροπία. Πρέπει να δούμε και εκεί τι γίνεται. Νομίζω ότι η συζήτηση αφορά τελικά τα μεγάλα αεροδρόμια ε, με πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών. Γενικά, Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε την αύξηση του ανταγωνισμού. Αν κοιτάξουμε λοιπόν και την νομοθετική παρέμβαση, όταν έχει τα συμβατικέ υποχρέωσει ανάμεσα σε ένα πελάτη και μια εταιρεία, αυτό εξασφαλίζει τον ανταγωνισμό. Και αν δείτε τον ε, πελάτη, εταιρείε ε, πάροχη υπηρεσιών, ε, η πίεση του πελάτη λειτουργεί ούτω ώστε ε, υπάρχει υπηρεσιών εδάφους να κάνουν τη δουλειά τους. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Τι πρέπει να νομοθετούμε, πού πρέπει να νομοθετούμε, ποιος είναι ο ρόλος της Κομισιόν. Πρέπει να λειτουργήσουμε με λογική, ούτω ώστε να μην έχουμε τεράστιες νομοθετικές διαδικασίες, όλα να είναι επιτακτικά ε, καθορισμένα για όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι και αυτό είναι ιδανική λύση. Ε, εκ μέρους της ECR θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζασάντα και νομίζω ότι αυτή η γενική προσέγγιση του Συμβουλίου είναι η σωστή. Φυσικά υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια κράτη-μέλη, πρέπει να επιληθούν, αλλά συνολικά η προσέγγιση του Συμβουλίου είναι καλή και ευχαριστώ τον ε, εισηγητή. Λοιπόν, Δύο λεπτά για το μακρύ κατάλογο των ε, ομιλητών που έχω. Η κυρία Ντεβεράκ είναι η πρώτη και μετά θα μιλήσει και το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Εξήγησα τη θέση της ε, Κομισιόν. Η θέση της Κομισιόν μάλλον για, τις, ε, για τους ενδιάμεσους σταθμούς είναι σωστή. σήμερα η αγορά είναι αρκετά όρημη για να ανοίξει περαιτέρω. Ε, χαιρετούμε τις ε, προσπάθειες των αεροδρομίων εδώ και 10 χρόνια για να ανοίξουν στην απελευθέρωση. Ε, κάποια αεροδρόμια όμως ε, καθυστερούν σε αυτόν τον τομέα ε, και δεν έχουν να προσφέρουν μια πλειάδα υπηρεσιών στους χρήστες τους. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την, τον κύριο Ζασάντα για τη δουλειά του, για το σχέδιο έκθεση που συζητάμε σήμερα. Ε, είναι αντικείμενο συμβασμού, αν το συγκρίνουμε με τις προτάσεις που έγιναν στο έγγραφο εργασίας που μοιράστηκε πριν από λίγους μήνες. Ε, είναι σημαντικό να μην διευρύνουμε την έννοια της, του αυτοχειρισμού. Πρέπει να διατηρήσουμε την διαταξή που απαγορεύει την υπεργολαβία. Ε, εδώ συμφωνώ με το τελικό κείμενο του συναδέλφου. ό,τι αφορά την πρόταση που κάνουμε να αυξήσουμε τον ελάχιστο αριθμό των παρόχων σε 4 αντί για τρία για τα μεγάλα αεροδρόμια, ε, μέχρι πριν από λίγο είχα κάποιες επιφυλάξεις. Ε, και αν τελικά χρειάζεται αυτό για να ανοίξει περισσότερο η αγορά ε, σε αυτά τα λίγα αεροδρόμια που μοιάζουν με γαλατικά χωριά, γιατί όχι. Το θέμα είναι να προσφέρουμε στους χρήστες ε, μια πλειάδα υπηρεσιών, λαμβάνοντας, στους χρήστες, λαμβάνοντας υπόψη και το χώρο των αεροδρομίων. πολλά αεροδρόμια μπόρεσαν να προσαρμοστούν στην έλευση αυτών των νέων παρόχων. Το άνοιγμα επίσης δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ε, ποιότητα της υπηρεσία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ γιατί συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια Ασφάλεια ενεργητική και παθητική των αεροδρομίων. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον συνάδελφο, να βάλουμε στο παράρτημα ένα γενικό πλαίσιο ε, κανόνων ε, ποιότητα. Πέρα από τον όρο πάροχη, είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που έχουν πολλές διοικητικέ υποχρεώσει και αμφισβητώ την ανάγκη να αυξήσουμε την ανάγκη υποβολής εκθέσεων προς την Κομισιόν. Έχω χρόνο να μπω και για... στα θέματα της κρίσης. Όχι, δεν έχετε. Σας το λέω καθαρά και ανοιχτά. Θα αρχίσω να σας χρονομετρώ. Κυρία Γουίλς, ζητώ συγγνώμη σας ξέχασα, δεν είσαστε στον κατάλογο των σκιωδών μιλητών, εκπροσωπείτε την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η διάνοιξη της αγοράς μέχρι τώρα οδήγησε σε μείωση της ποιότητας στις υπηρεσίες εδάφους και ε, μείωση το μισθό μέχρι 20%. Ε, ε, απασχολούμενοι εκεί δεν μπορούν να επιβιώσουν και ο ανταγωνισμός στην αγορά θα πρέπει να είναι ε, προσανατολισμένο στην ποιότητα της προσφοράς και όχι στο χαμηλότερο κόστος προσωπικού. Για μένα τα εξής κριτήρια είναι ουσιώδου σημασίας. Οι αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις, συμφωνώ με τον κύριο Φλέκενστάιν, ποιοτικέ προδιαγραφές για την κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση, να απαγορεύονται οι υπεργολαβίες και να εξασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας τουλάχιστον με τις ίδιες συνθήκες όταν αλλάζει ο πάροχος. Ε, εκτός αυτού είμαι κατά της αναγκαστικής ε, διάκρισης ε, της νομικής από τις εταιρείες των αεροδρομίων θα πρέπει να υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες και σημαντική βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης των εργαζομένων για να τεθούν όλα αυτά σε ισχύ. Με τρομάζει το γεγονός ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι, λέει, αρκετά φιλόδοξη για τον εισηγητή. Με ε, ανταγωνισμό και περαιτέρω απελευθέρωση θα πέσουν οι τιμές και ε, υποτίθεται θα αυξηθεί η ποιότητα. Έτσι τα φαντάζεται ο εισηγητής. Και γι' αυτό θέλει ε, τον ελάχιστο αριθμό των παρόχων στα μεγάλα αεροδρόμια το αυξήσει κατά ένα, από τρεις σε τέσσερις. Και να υπάρχουν και υπεργολαβίες. Και έτσι, ε, οι εταιρείε που είναι στον ίδιο όμιλο θα μπορούν να αναθέτουν μεταξύ τους τις υπηρεσίες. Την περασμένη εβδομάδα ήρθαν τα αποτελέσματα μιας μελέτης ε, ε, που έγινε ε, από συνδικάτα και διαφερομένους και δείχνει ότι ε, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας και ε, τελικά σε ανασφάλιστη εργασία σε αυτές τις υπηρεσίες εδάφους. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις μεταφορές Έκανε μια δράση αρχές Ιουλίου ε, πάνω στις κάρτες επιβίβασης και γράφει stop στην απελευθέρωση γιατί ε, ε, θα επιδεινώσει την κατάσταση. Εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι μαζί με τα συνδικάτα. Θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη και όχι την Ευρώπη των dumping των μισών. Λοιπόν, τώρα θα βάλω ρολόι να το βλέπετε. Ο κύριος Λάιχφριτ, δύο λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κλίντς Αναφέρθηκε στην ελευθερία του επιχειρήν. Εγώ θα το πω αλλιώ. Εμείς το λέμε αυτή η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Και διαπιστώνω εδώ και πώς φαντάζομαι εγώ ε, τον κλάδο αυτόν. Μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα εταιρείε εταιρείες που θα προσδιογιώνονται, με βάση τα συμφέροντά τους. Και οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν από ποιο αεροδρόμιο θα φύγουν. Αυτό είναι σαφές σχετικά. Και κανείς δεν διαμαρτύρεται που ισχύει. Επίσης φαντάζομαι ότι τα αεροδρόμια μπορούν να προσφέρουν ό,τι θέλουν να προσφέρουν. Και αυτό ανήκει σε μια κοινωνική ελεύθερη αγορά. Και ακούμε τους υπαλλήλους, τις κυρίες και τους κυρίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ε, επίτροπο, τον αρμόδιο, που ενδιαφέρεται λιγότερο για να ρυθμίσει τα πράγματα και περισσότερο για να περάσει την ιδεολογία του, αν του αφήσουμε ελεύθερους, θα αναγκάσουν τα αεροδρόμια πόσους ε, παρόχους μπορούν να λειτουργούν εκεί και με ποιες προϋποθέσεις. Αυτή είναι η ελευθερία της αγοράς. Αυτό είναι καταναγκασμό. Πρώτον, δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα, ούτε την εξυπηρετεί, δεν εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντα των εργαζομένων και τελικά ε, ούτε τα συμφέροντα των επιβατών. Το πολύ πολύ ε, βοηθάει κάποιους που θέλουν να βγάλουν χοντρά λεφτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε μία κατάσταση που δεν ε, την αντιλαμβάνονται ως ιδεώδη οι πολίτες και ιδιαίτερα εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Και εμείς δεν έχουμε άλλη δουλειά από το να επιδεινώνουμε περαιτέρω την κατάσταση. Δεν είναι καλά αυτά. Και κύριε Σασάντα, το ξέρω, έχετε και άλλα ενδιαφέροντα ίσως και συμφέροντα, αλλά μην σκέφτεστε μόνο την οικονομική πολιτική και τα οράματά σας που μπορεί να είναι σπουδαία για σας. Σκεφτείτε και τους ε, εργαζομένους, άνδρες και γυναίκες, επιβάτες άνδρες και γυναίκες, γιατί αυτούς σε καμία περίπτωση δεν τους εξυπηρετεί η δική σας πρόταση. Ο κύριος Γκρό, Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα ε, και εγώ να ευχαριστήσω τον Άρτουρ. Γιατί μιλάνε τόσοι Γερμανοί. Πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό το θέμα μιλάνε την ίδια γλώσσα βέβαια, αλλά όχι με την ίδια φωνή. Ε, δεν θα είναι εύκολο για τον κύριο Σασάντα να καταλήξει συμβιβασμό. Θα πρέπει να ε, οδηγήσουμε τη συζήτηση εκεί που ανήκει. Ποιος είναι ο στόχος αν θέλουμε να αυξήσουμε ε, τον αριθμό των επιβατών, ε, δεν είναι απάντηση να έχουμε περισσότερους παρόχους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ασφάλεια των πτήσεων. Εάν θέλουμε λοιπόν, όχι αυτό, αλλά να οργανώσουμε την αγορά, θα πρέπει να προέχει η ποιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μειώνει την ποιότητα όταν είναι περισσότεροι οι πάροχοι γιατί τότε κάθε αεροπορική εταιρεία θα επιλέξει τον καλύτερο για να παρέχει την καλύτερη ποιότητα. Γιατί ποιότητα σημαίνει και ασφάλεια. Γι' αυτό το στοιχείο τη ασφαλεία θα πρέπει να συνυπολογίζεται. Για την εσωμάτωση, τον νομικό διαχωρισμό, την αυτοδιαχείριση των αεροδρομίων, τα έχουμε πει αυτά. Ε, θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε και ω προ την οικονομικότητα. Το τελευταίο έχει να κάνει με την με τις με, το χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, επεκτείνεται ένα αεροδρόμιο. Εξαγγέλει ότι θέλει ένα νέο πάροχο, αλλά μετά λέει δεν έχω χώρο. Μα ε, τι θέλει ο επιβάτης, ποιότητα. Σήμερα υπάρχει μεν ποιότητα, αλλά όχι παντού. Ο, ο επιβάτης δεν θέλει κατά ανάγκη φτηνότερες τιμές, θέλει καλύτερη ποιότητα και το τονίζω αυτό και ένα τελευταίο. Το κοινωνικό dumping δεν είναι του παρόντος ε, Κανονικά μέχρι σήμερα το ορίζει η κάθε περιφέρεια και το κάθε κράτος το ίδιο, μπορούν να το κάνουν και τα αεροδρόμια. Ο κύριος Χαντράου για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Σε σχέση με το σημείωμα για τη συζήτηση έχει κάνει βήματα προς τα μπρος, αλλά παραμένουν κάποια σημεία τριβή. Τα έχουν πει ήδη συνάδελφοι από την πολιτική μου ομάδα. Βεβαίω έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, η συζήτηση για τον αριθμό των παρόχων. Εμεί τι φρονούμε φτάνουν οι δύο τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα να το καθορίζει το κάθε κράτος μέλος αν χρειάζεται περισσότερο ή όχι. Ωραίο αυτό. Δεν χρειάζεται να το ρυθμίσουμε ευρωπαϊκά αυτό το θέμα. Εγώ δεν είμαι ε, του να, ε, κατά του υπάρχει μια ε, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών εδάφους από το ίδιο το αεροδρόμιο. Υπάρχουν αεροδρόμια που δουλεύουν νύχτα, α πούμε, και το καλύτερο είναι μόνο τους να τα ρυθμίζουν αυτά τα θέματα και τις ε, ε υπηρεσίες ε, ε, αυτό που θεωρώ θετικό στην έκθεση είναι η πρόταση για τα ποιοτικά κριτήρια. Βεβαίω, θα τα κοιτάξουμε με την ησυχία μας, αλλά καλό είναι να βάλουμε και τέτοια κριτήρια. Και η προσοχή που δίνεται για ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα και άτομα με αναπηρίες και την υποχρέωση ενημέρωσης στα ίδια τα αεροδρόμια και τους χρήστες. Τώρα κάνουμε μια άσκηση στην Επιτροπή ε, Μεταφορών, αλλά δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε χωριστά από αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι μας στην Κοινωνική Επιτροπή, διότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον τομέα αυτό να κάνουμε πρόοδο και συγκεκριμένα όταν πρόκειται για την πρόσληψη υπαλλήλων όταν χάνονται οι συμβάσεις και την κερδίζουν κάποιοι άλλοι, άλλες εταιρείες, δεν θα πρέπει να είναι αυτό εις βάρος των εργαζομένων ε, και να την πληρώνουν αυτοί. Κατά τα άλλα, αν δούμε και τα κοινωνικά, θα είναι καλή έκθεση. Για τον αριθμό λοιπόν των παρόχων ε, σημαντική συζήτηση και κατά τα άλλα, από αυτό θα εξαρτηθεί τελικά η στάση μας αν θα υποστηρίξουμε την έκθεση ή όχι. Ευχαριστώ κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στον κύριο Σασάντα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά και καλές προτάσεις. Προσωπικά για μένα δεν γίνονται σεβαστοί όμως κάποιοι βασικοί κανόνες και συμφωνούν πολλοί σε αυτό, ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να θέτουν μόνο ένα πλαίσιο και από εκεί και πέρα να ε, λαμβάνονται υπόψη περισσότερο οι εθνικές ε, συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Συμφωνώ για την ποιότητα, για την ασφάλεια, να ρυθμίζονται αυτά πανευρωπαϊκά. Αλλά την απόφαση για την περαιτέρω απελευθέρωση θα πρέπει να την παίρνουμε όσο γίνεται πιο κοντά στο πολίτη. Βλέπε επικουρικότητα στα κράτη-μέλη. Και για την αναλογικότητα. Πιστεύω ότι το παρατραβάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με την οδηγία 96. Εντάξει, διάνοιξη αγορά. Μα δεν υπάρχει μονοπωλιακή θέση που θέλω. Είμαι κατά το μονοπωλίο, ρε παρόδο να το πω, αλλά είμαι και κατά μια περαιτέρω απελευθέρωση για λόγου αμυγό ιδεολογικού. Και πιστεύω και εδώ ότι περαιτέρω διάνοιξη ε, είναι προβληματική. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Πολλέ δυσκολίε και στον κοινωνικό τομέα αλλά και στον οικονομικό. Πιστεύω ότι αν ανοίξει κι άλλο η αγορά δεν θα έχουμε προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό πρέπει να σας πω την προσωπική μου άποψη ότι πρώτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ε, απορριφθεί και να έχουμε οδικία πλαίσιο και όχι κανονισμό και να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη με βάση την επικουρικότητα το δρόμο που θα ακολουθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπαχ. Ο κύριος Ντεμπάκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε ε, και υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Εδώ συμφωνούμε όλοι ότι για τις υπηρεσίες εδάφους το status quo δεν είναι εναλλακτική λύση ε, και χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή. Ε, γι' αυτό χαιρόμαστε για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπε ο κύριος Λάιχφριτ ότι κάθε αγορά χρειάζεται κανόνες, βασικούς κανόνες. Και ένας από αυτούς είναι ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση ε, με τρόπο διαφανή και ειλικρινή. Αυτό προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω λοιπόν και να χαρώ. Αυτός ο κλάδος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας κανονικός κλάδος της οικονομίας που χρειάζεται και άλλη απελευθέρωση, ελεύθερο ανταγωνισμό και αυτό θα αυξήσει την ποιότητα ε, των παροχωμένων υπηρεσιών για τους ε, επιβάτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί ε, το νομικό διαχωρισμό τον έχει κάνει λειτουργικό διαχωρισμό. Ε, έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση και στο σιδηρόδρομο και χρησιμοποιούνται διάφορες προφάσεις. Όχι, εγώ θέλω να υπάρχει και ε, νομοθετικός διαχωρισμός. Και τώρα η βάση της συζήτησης έχει να κάνει με τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κατεξουδότηση πράξης και εγώ θα ήθελα να υπάρξει περαιτέρω εναρμόνιση γιατί κάθε επιβάτη στην Ευρώπη περιμένει τις ίδιες ποιοτικέ προδιαγραφές. Και σε ό,τι αφορά την απασχόληση έχω δει τα πιο μυστήρια πράγματα. Μα είναι ήδη προστατευόμενος ο τομέας αυτός γιατί χρειάζεται περισσότερη προστασία. Θα πρέπει να είναι μια συνήθις αγορά με τις κανονικές συνθήκες ε, που επικρατούν σε όλους τους κλάδους της αγοράς. Και θα περιμένω και τις προτάσεις Επιτροπής Απασχόλησης για να δούμε πώς μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε στη δική μας έκθεση. Κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ βλέπω μια σειρά μεγάλων δυσκολιών και ανοιχτών ζητημάτων αρχής γενομένης από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε από λάθο αφετηρία και ποτέ δεν έλαβε υπόψη σοβαρά όλες ε, τις προϋποθέσεις. Ένα κράτος μέλος που θέλει σήμερα να απελευθερώσει μπορεί να το κάνει. Δεν του χρειάζεται αυτός ο κανονισμός. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Και πιστεύω ότι εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν ρυθμισμένη αγορά έχουν και λόγους που τις έχουν αυτές τις αγορές. Λειτουργούν καλά τα αεροδρόμια με καλύτερες υπηρεσίες από κάποιες άλλες χώρες και αεροδρόμια που είναι τελείως ελεύθερα. Κάτι άλλο που δεν έχω καταλάβει είναι η σχέση μεταξύ του ωραρίου των εργαζομένων ε, σε, χώρες, σε ώρες εχμής και ώρες ε, μη εχμής. Αυτό ονομάζεται παραγωγικότητα ε, των εργαζομένων. Όταν είναι περισσότεροι υπάροχοι αλλά οι ίδιοι νεκροί χώροι, νεκρές περίοδοι, δεν βοηθάει αυτό στην αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του αεροδρομίου. Θα ήθελα να δούμε ποια είναι η ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν ε, κάποιες ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, κάποιες υπηρεσίες που παρέχει το αεροδρόμιο και οι υπόλοιπε ε, είναι στο 20% της αγοράς. Ε, εκεί που είναι τελείως ανοιχτή η αγορά, είτε αυτό το Λονδίνο είτε το Άμστερνταμ, η ποιότητα και η ακρίβεια στο χρόνο δεν είναι καλύτερη από ό,τι στη Φραγκφούρτη, για παράδειγμα. Ε, και η ανάπτυξη και η μεγέθυνση της οικονομίας δεν θα ε, αλλάξει τα μερίδια στην αγορά. Είναι θέμα ασφαλείας και δεν θα πρέπει να κάνουμε πειράματα εδώ. Και ερχόμαι στο τέλος. Ε, δεν μας χρειάζεται αυτός ο κανονισμός και μπορούμε να απορρίψουμε, να επαναπέψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση στο σύνολό της. Ο κύριος Πίρκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Ποιο είναι ο στόχος μας. Τρεις είναι οι στόχοι τουλάχιστον. Οι επιβάτες και οι αερομεταφορείς θα πρέπει να ε, και θέλουν γρήγορη και ασφαλή ε, υπηρεσία εδάφους με χαμηλό κόστος αλλά με καλή δουλειά και ε, όχι κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά σεβασμό στους εργαζομένους. Θέλω να προτείνω τα εξής. Πρώτον, Η ισχύουσα οδηγία δίνει τη δυνατότητα για την απελευθέρωση της αγοράς. Όταν λένε τουλάχιστον δύο πάροχοι, όταν λένε τουλάχιστον δύο, προφανώς μπορεί να είναι και περισσότεροι από δύο. Δεν χρειάζεται νέα ρύθμιση ή αλλαγή ή καθορισμός ε, συγκεκριμένου αριθμού παρόχων. Στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε καλύτερες ε, διαδικασίες δημοσίων διαγωνισμών με μεγαλύτερη διαφάνεια. Στη συνέχεια, ελάχιστες προδιαγραφές, ποιοτικέ, πανευρωπαϊκά, ναι. Να μην αποφασίζει το κάθε αεροδρόμιο ή κάθε χώρα ε, τι θα ισχύει. Ε, και για να μειώσουμε το κόστος θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, εμείς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να κάνει ό,τι μπορεί για να υλοποιηθεί ε, ε, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ε, ουρανός. Αυτή η πρόταση που κάνει τώρα για κανονισμό δεν χρειάζεται για να επιτύχουμε τους στόχους που επιθυμούμε. Ευχαριστώ κύριε Πίρκερ. Πριν δώσω λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω δύο λόγια εγώ. Και εγώ θα εστιαστώ στην ποιότητα για τις ε, πηγή εξυπηρέτηση. Συμφωνώ ότι βέβαια η οδηγία πηγαίνει πέρα από αυτό, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ένα θέμα. Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται στους επιβάτες έχει μειωθεί, έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής, ε, χάνονται αποσκευές. Ε, όλοι φαντάζομαι έχουμε τέτοιες εμπειρίες προσωπικές από ε, κάποιον πάροχο ο οποίος έχασε την βαλίτσα μας επειδή ήταν μακριά το αεροπλάνο παρκαρισμένο και μας ε, ακούμε και από μιλητές εδώ να μας λένε ότι στα αεροδρόμια του Φραγκφούρτης τα λεωφορεία πέφτουν το απανοστάλο. Λοιπόν υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε όλα τα αεροδρόμια. Αλλά για εμένα θα πρέπει να εστιάσουμε στο πρόβλημα της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχεται. Ακούμε να λένε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα των αεροπορικών εταιριών οι οποίες θα έρθουν σε επαφή με τις εταιρείες που παρέχουν εξυπηρέτηση. Αλλά εάν οι ε, ε, αεροπορικέ εταιρείε προσπαθούν να πάρουν όλο και πιο χαμηλή τιμή από αυτές τις ε, εταιρείε η πηγε εξυπηρετησης ειναι αναποφευκτο οτι η ποιοτητα θα μειώνεται και θα γίνεται όλο και χειρότερη. Και σε αυτό θα έπρεπε να, με αυτό θα έπρεπε να ασχοληθούμε. Όπως είπε και ο κ. Κλίντ, γιατί ασχολείται η Επιτροπή απασχόληση. Για... όλες οι πολιτικέ ομάδε, συμπεριλαμβανομένε και τη δική σα. ε, έχουν μία άποψη σε σχέση με τον κανονισμό 50, του άρθρου 50 του κανονισμού. Η δικιά μου άποψη δεν ξέρετε, αλλά είναι μειοψηφία. Τώρα, ε, δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Merci, le Κυρία Μέη, ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω το έργο που έχετε επιτελέσει ως Επιτροπή συνολικά στο θέμα αυτής της έκθεσης. Για να ανταπαντήσω στον κύριο Κλίντ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι πλήρως δεσμευμένη και προσπαθεί να προωθήσει τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Είναι ζήτημα ανταγωνισμού, δίκαιου και ισότιμου και σε σχέση επίσης με τους ε, εταίρους μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ανακοίνωση της Επιτροπής ε, στις 27 Σεπτεμβρίου σε σχέση με το θέμα. Τώρα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. λόγω της συνθήκης, εμείς οφείλουμε να είμαστε ουδέτεροι στο θέμα και δεν μπορούμε να επέμβουμε. Όσον αφορά τη βοήθεια στους ανάμεσους σταθμού και την, αναφορά, την έκθεση του κ. Ζασάντα, ο οποίο ε, αναφέρεται στην ισορροπία που προσπαθεί να επιτύχει η Επιτροπή μεταξύ του ανοίγματο της αγοράς και της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων, που επίσης συνδέονται και με την ποιότητα των υπηρεσιών. Η θέση μας είναι εξή. Ε, καλωσορίζουμε την δουλειά που έχει γίνει για τους ελάχιστους κανόνες ποιότητας. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συζητούνται αυτά τα ζητήματα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μην ε, υπάρχουν πολλαπλά και διαφορετικά ε, πρότυπα στο τοπικό επίπεδο, κάτι που θα δυσκολέψει την λειτουργία των αεροπορικών εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα πρότυπα ποιότητα πρέπει να συμφωνούνται σε, ευρωπαϊκό, επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, θεωρούμε την εισήγηση του κυρίου Ζασάντα θετική βάση για την επικυρωποίηση της οδηγίας ε, του 2007-96 σας 996 μας είχε ζητηθεί μία εις ε, μελέτη για την εξυπηρέτηση των ενδιάμεσων σταθμών και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματική και ποιοτική. Και με αυτήν την πρόταση της Επιτροπής προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο που μας είχε ανατεθεί. Δηλαδή, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους επιβάτες. Σας ευχαριστώ. Ζασάντα, μήπως θα θέλατε σύντομα να προσθέσετε κάτι. Ναι, πολύ σύντομος θα είμαι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που ε, κάνατε σχόλια και εξετάσατε με προσοχή το έγγραφο που παρουσίασα και που παρουσία... επίσης εντοπίσατε το γεγονό ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για την απελευθέρωση των... της αγοράς και στα αεροδρόμια. Το ζήτημα εδώ είναι η εισαγωγή ελάχιστων προτύπων ποιότητας στα αεροδρόμια έτσι ώστε όλοι οι επιβάτες να έχουν την ίδια ε, να απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης εκείνη για την οποία πλήρωσαν εν τέλει. Σήμερα ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μας λένε ότι δεν είναι δυνατόν να εξαναγκάσουν τις ε, εταιρείες πήγες εξυπηρέτησης να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες γιατί έχουν μόνο δύο εταιρείες και οι δύο παρέχουν την ίδια ποιότητα και καμία από τις δύο δεν ενδιαφέρεται να αυξήσει και να βελτιώσει την ποιότητά της. Να γιατί έχουμε παρουσιάσει αυτήν την πρόταση έτσι ώστε να αναγκαστούν οι εταιρείες να ανταγωνιστούν η μία την άλλη και να ανταγωνιστούν στη βάση της ποιότητας και μόνο. Η ποιότητα η οποία θα ε, καθορίζεται από τα αεροδρόμια, γιατί θεωρώ ότι τα αεροδρόμια, το κάθε αεροδρόμιο γνωρίζει καλύτερα ποιος θα είναι ο ελάχιστος χρόνος μεταφοράς μιας ε, αποσκευής από το αεροπλάνο μέχρι το τερματικό σταθμό κτλ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν θα καταφέρει να γνωρίζει καλύτερα και να υπολογίσει από τις Βρυξέλλες ποιο θα πρέπει να είναι ο χρόνος μεταφοράς των αποσκευών. Ε, όλες, όλες αυτές τις παραμέτρους δεν θα μπορέσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις ε, ε, αποφασίσει καλύτερα από τα ίδια τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια λοιπόν θα υιοθετούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητα και μετά αυτά θα εγκρίνονται από τι αρμόδιε αρχέ στα κράτη-μέλη. Έτσι θα αναγκαστούν οι εταιρείε παροχή πηγή εξυπηρέτηση να αυξήσουν την ποιότητά του, να παράσχουν ε, καλύτερη ποιότητα υπηρεσίε στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Σα ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ζασάντα. Φαίνεται πόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για την έκθεσή σας από τον τεράστιο κατάλογο ομιλητών που συγκέντρωσα. Ε, σας εύχομαι καλή τύχη τώρα που θα εργαστείτε με τους κοιόδης συζητητές. 26 Σεπτεμβρίου είναι το, η προθεσμία για τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να έχουμε τόσο αυστηρή διαδικασία και με την επόμενο μέρος της ε, εισήγηση που αφορά στον θόρυβο. κύριος Λάιχτριχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. μια ωραία ταινία, μπορούμε να τη δείξουμε. Ε, τώρα προκαλείτε την τύχη σας κύριε Λάιχφριτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταφέραμε τώρα να φτιάξουμε μια έκθεση μια πρόταση ε, για την έκθεση για το θόρυβο. Και έχουμε τώρα την ευκαιρία ε, να παρουσιάσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία. Ε, το μεγαλύτερο θέμα ποιο ήταν. Τι γίνεται σήμερα στα κράτη-μέλη τηρούν τα διεθνή πρότυπα για την προστασία από το θόρυβο. Ε, χρειάζεται βελτίωση. Αυτό ήταν και ε, εκείνο που όθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτή την πρόταση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και πραγματικά το κατανοούμε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Στις συζητήσεις μας όμως είχαμε ένα μεγάλο σημείο τριβής. Τι θα γίνει με το άρθρο 10. Το άρθρο 10 της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε, ε, έχει ιδιοποιηθεί το δικαίωμα να ελέγχει ε, τα όσα ισχύουν στα κράτη-μέλη, να τα εγκρίνει, να τα απορρίπτει. Μα πέρα από τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλα συμφέροντα και κάποιοι υπερατλαντικοί εταίροι μας συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση αλλά κατέληξα στο εξής αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Ένας λογικός συμβιβασμός θα πρέπει να έχει ως εξής. Η πραγματική απάντηση και απόφαση τελικά θα πρέπει να λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. στο βαθμό που έχει άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνεται και αυτή η υπόψη. Αλλά από την άλλη δεν θα πρέπει να έχει μια ύπατη αρχή στις Βρυξέλλες τη δυνατότητα κατάργησης ή ακύρωσης τοπικών αποφάσεων. Υπάρχει διαδικασία έκτακτη στη γενική ε, διαδικασία προσφυγής επί παραλήψη. Ε, το έχει αυτό το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό θα πρέπει να αρκεί. Ιδιαίτερα γιατί με αυτό το κανόνα, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, δεν λύνεται το εξής πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτο το κανονα οπως προτεινεται απο την ευρωπαικη επιτροπη δεν λυνεται το εξή προβλημα τι γινεται με αποφασεις που δεν λαμβάνονται από κρατικές αρχές, κανόνες δικαίου δηλαδή, αλλά ε, τι γίνεται με λύσεις για την προστασία ε, από θόρυβο που έχουν γίνει μετά από μια διαδικασία διαμεσολάβησης και συνδιαλλαγής μεταξύ των ενδιαφερμένων φορέων. Ε, υπάρχουν ιστορίες που διαρκούν έτη πολλά και διαπραγματεύονται αεροδρόμια με γείτονε, με φορείς, με οργανώσεις και τελικά βγαίνει ένα αποτέλεσμα πάνω κάτω αποδεκτό από όλους αυτό μπορεί να έρθει μια αρχή των Βρυξελών και να το καταργήσει, δεν μπορώ να το φανταστώ. Και ε, γι' αυτό έκανα και την πρότασή μου για την έκθεση. Επιπλέον, προσπάθησα να ξαναβρω ένα ορισμό που θεωρώ σημαντικό. Η λεγόμενη ισορροπημένη προσέγγιση πάντα γινόταν ε, λόγος για το κόστος, ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένο το κόστος. Εγώ θα πρέπει ε, να σας πω ότι μιλώ γενικότερα για αποτελεσματικότητα, όχι μόνο το κόστος και προστασία της δημόσιας υγείας και αποτελεσματική προστασία από το θόρυβο, αποτελεσματικά μέτρα. Δηλαδή αυτή η έννοια της αποτελεσματικότητας είναι πολύ ευρύτερη και γενικότερη από το αμυγές οικονομικό κόστος. Αυτά σε γενικές γραμμές τα βασικότερα στοιχεία που άλλαξαν και από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι άλλο που ήρθε να προσθεθεί. Κοίταξε και τους τύπους των αεροσκαφών και Νομίζω ότι οι οριακές τιμές που ισχύουν σήμερα είναι εντάξει. Αν θέλετε μια προθεσμία που μπορούμε ε, να την ορίσουμε, μπορούμε να περάσουμε από το 8 στο 10. Ε, σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξη, πράξης, μπορεί να γίνει αυτό σε αμυγός όμως ε, τεχνικά ζητήματα. αλλά οτιδήποτε μπορεί να έχει πολιτικές συνέπειες, όπως οι οριακές τιμές εκπομπών θορύβου κτλ. δεν ε, προσφέρεται η κατεξουσιοδότηση πράξη για να λύνεται αυτό. Θα πρέπει στην απόφαση να συμμετέχει άμεσα το κοινοβούλιο. Εμείς πρέπει να τα αποφασίζουμε αυτά που είμαστε πρόσωποι των πολιτών στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι αντέδρασαν πάρα πολύ από παντού από την Ευρώπη, πάρα πολλά email πήρα που βεβαίως με βοήθησαν πολύ και με υποστήριξαν και πολλοί, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και μελήματα και ανησυχίες που δεν μπόρεσα να συμφωνήσω. Ας πούμε, δεν προβλεπόταν σε αυτό τον κανονισμό ε, να βάλω συγκεκριμένες οριακές τιμές, ούτε η Κομισιόν το ζητάει, ούτε εμείς στην έκθεσή μας. Δεν ήταν αντικείμενο αυτής της πρότασης, ούτε νόημα. Επίσης δεν μπορούμε να αλλάξουμε διεθνείς συμφωνίες ούτε να αλλάξουμε την ισορροπημένη προσέγγιση. Είναι μια διεθνής συμφωνία και δεν μπορεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης μονομερός να την αλλάξει. Και αυτό λοιπόν είναι σαφές. Αλλά γενικά, αλλάζοντας αυτό το αποτελεσματικό ως προς το κόστος, να το κάνουμε γενικότερα αποτελεσματικό, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και τέτοια μελήματα. Ας πούμε θέλουμε στο μέλλον οι Ευρωπαίοι να μπορούν να κοιμούνται πιο ήσυχα και καλύτερα, αλλά να τηρούμε και τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτή είναι η απαραίτητη συμβαστική πρόταση και περιμένω με χαρά να ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων με τους οποίους έχουμε αγαστή συνεργασία από τώρα, έτσι και και θέλω να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή για την καλή συνεργασία και τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ και εγώ ανταποδίδω. Όντως, οι κατεξουδότητες πράξης, όπως είπατε και εσείς, δεν προσφέρονται ε, για τις οριακές τιμέ και για θέματα τέτοια πολιτικά. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερο λόγο επί της ουσίας, όχι των τεχνικών θεμάτων. Συμφωνώ πάρα πολύ με το άρθρο 10 και τη νέα διατύπωση του, της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να μπούμε ακριβώς σε αυτό το δρόμο για να μπορούμε και να ε, αφήνουμε τις ε, αποφάσεις να λαμβάνονται επί τόπου. Συμφωνώ με αυτό που είπατε εσείς. Ε, σε ό,τι ε, αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για τα αεροσκάφη, υιοθετείτε αυτό που πρότεινε το Συμβούλιο. Θα μπορούσα να συμφωνήσω κι εγώ. Είναι ένα σημείο το οποίο εγγράφεται στα πλαίσια του συμβιβασμού και αυτό και μπορεί να περάσει. Εγώ να δείτε email που πήρα. Και οι υπόλοιποι φαντάζομαι για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την ποιότητα ζωής. Βέβαια, κατανοώ την επιθυμία των ενδιαφερομένων, γιατί αυτοί που γράφουν ε, μένουν κοντά σε αεροδρόμι. Αλλά προβληματίζομαι. Ε, ποιες θα ήταν οι μέθοδοι μέτρησης για να αποδείξει κανείς κάτι σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Πώς επηρεάζει ο θόρυβος στην υγεία ε, έχει αυτό αποδειχθεί, Εάν όχι, το μόνο που βλέπω είναι να ανοίγει μια τεράστια αγορά για τους δικηγόρους ε, που θα δραστηριοποιηθούν. Και θα μπορούσε αυτό να βλάψει ή να απειλήσει κάποια αποτελέσματα ε, διαδικασιών συνδιαλλαγής και διαμεσολάβησης. Εδώ χρειάζεται συζήτηση ακόμα. Συμφωνούμε να περιορίσουμε το θόρυβο, αυτό είναι ο στόχος μας, αλλά να το κοιτάξουμε. Και πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Για τον νέο ορισμό του τι εστί αποτελεσματικότητα ε, ως προς το κόστος, ή μια γενικότερη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ίσως αυτό χρειάζεται να συζητηθεί ακόμα Πάντως στον κανονισμό να το ορίσουμε τι σημαίνει αυτό περιορισμός και ε, αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος σε σχέση με το γενικότερο, το overall cost efficiency. Γιατί και πάλι θα τρίβουν τα χέρια τους οι δικηγόροι. αλλά τα σημαντικότερα σας είπα είναι το θέματα του άρθρου 10. Συμφωνούμε μαζί σας από πλευρά του ΕΛΚ. Ε, είμαστε στον ίδιο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας. Κύριε Βέρνε, συζητώ συγγνώμη από την Επιτροπή Περιφερειών. Έπρεπε να σας είχα δώσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Σίμψον, κύριε Λάιχφριτ. Ο θόρυβος είναι πολύ σημαντικό θέμα για τις περιφέρειες και τις πόλεις. Δεν είμαστε μόνο κοντά, ε, αλλά ε, και πολλές φορές είμαστε αρμόδιες αρχές ε, για να τα αποφασίσουμε. Η τεχνική εξέλιξη έχει περιορίσει σημαντικά το θόρυβο, αλλά ε, είναι γεγονός ότι ο θόρυβος ενοχλεί και περισσότερο κόσμο. Ο στόχος είναι να μειωθεί και να υπάρχει μια πιο ενιαία εφαρμογή των διαδικασιών στον περιορισμό της λειτουργίας των αεροδρομίων. Επίσης, κύριε Λάιφριτ, ε, βλέπουμε το πρόβλημα κυρίως σε αεροπλάνα που μεταφέρουν ε, εμπορεύματα που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία μας, για τα αεροσκάφη που τηρούν τις προδιαγραφές οριακά. Ε, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε για μια τετραετία αυτό το 8 δεσιμπέλ και μετά να φτάσουμε στον αρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το περιορισμό της λειτουργίας είμαστε αυστηροί. Ζητήσαμε να διαγραφεί τελείως το άρθρο 10. Αλλά αυτό που προτείνετε εσείς μας φαίνεται πιο κομψό και τελικά ε, έχουμε τον ίδιο στόχο και αυτό που μας έκανε μας να ζητήσουμε διαγραφή. Και στις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης Διαφωνούμε. Άρα ζητούμε να διαγραφούν και τα άρθρα 11 και 12. Αλλά αν τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που προτείνει εσείς θα ήταν πολύ καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του κυρίου Τρεμόσα, ο οποίος λυπάται πάρα πολύ, αλλά κολλείεται, έχει τρεμερή διάλογο και με παρακάλεσε να μιλήσω εξ ονόματός του. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τον εισηγητή μα και ο κύριος Τρεμόζα λέει ότι σε γενικές γραμμές συμφωνεί, υποστηρίζει το έγγραφο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά γιατί μου τα έχει δώσει στα αγγλικά γραμμένα. So, um, the balance... Για την ισορροπημένη προσέγγιση, ο κύριος Τρεμόζα καλωσορίζει το ότι στο κείμενο της Κομισιόν δεν υπάρχει καμία αναφορά στους ε, περιβαλλοντικούς ε, στόχους ή στόχους υγείας, όπως στις συστάσεις του ΠΟΗ γιατί είναι τόσο πολύ φιλόδοξη αυτέ αυτές οι στάσεις που ακόμη και ο ΠΟΗ αναγνωρίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιούνται μόνο ω ε, κατεύθυνση, ως στόχος. Επίση, πιστεύει ότι δεν είναι σωστό το γεγονός ότι η εστίαση ε, μπαίνει σε ένα πυλώνα, δηλαδή στους περιορισμούς του λειτουργικού. Θέλω να πει ότι και άλλοι πυλώνες είναι σημαντικοί, τεχνολογική πρόοδος, ε, ε, σχεδιασμός ε, των διαδικασιών, χρήση γης κτλ. Για την, σε εποχή οικονομικής κρίσης θα πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές πριν τιμωρήσουμε τον κλάδο και τους επιχειρηματίες. κάτι μπορεί να μας οδηγήσει σε απαγορεύσεις Κάτι τη νύχτα σε όλη την Ευρώπη. Ε, θα πρέπει και αυτό το οικονομικό κόστος να το βάλουμε, λάβουμε υπόψη μας για την Ευρώπη. Ως Γερμανίδα θέλω να πω ότι μου άρεσε η τροπολογία 38 του εισηγητή, γιατί λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγγύσει για την περίπτωση της Γερμανίας. το γερμανικό δικαστήριο, ας πούμε, αποφάσισε για απαγορεύσεις νυχτερινών πτήσεων ε, για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης πρόσφατα. για τα αεροσκάφη που μόνο οριακά συμμορφώνονται, ε, λέει ότι θα πρέπει να περιορίσουμε το, πέρα από τα 3 δεσιμπέλ στα 10. Ε, έτσι όμως μπορεί να ε, αυξηθούν οι εντάσεις μεταξύ το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ε, ΙΚΑΟ. Ε, η ΕΚΑΟ λέει τα κράτη-μέλη να μην ε, είναι υποχρεωτικό αυτό, να μην είναι υποχρεωτικά τα κεφάλαια 3 και κεφάλαια 4 για τα αεροσκάφη. Επίσης, ε, το όφελος για το περιβάλλον θα είναι πολύ υψηλό, αλλά το κόστος για τις εταιρείε θα είναι. Επίσης, και επίσης ο, τα, ο στόλος α321 δεν θα επηρεαστεί. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί κάποια ποσόστοση του, των αεροσκαφών, των περιφερειακών στόλου. Επομένως, για τα αεροσκάφη του κεφαλαίου 3-5 θα πρέπει να έχουμε μείον 8 DC. Ο κύριος Τρεμόζα λέει ότι είναι υπέρ της Βαρκελόνης πιστεύει στην επικουρικότητα, αλλά σε αυτήν την περίπτωση πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο η Κομισιόν μπορεί να ελέγχει εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων και υποτίθεται ότι αυτό είναι θετικό. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας ως Γερμανίδα που λέει ότι για τη Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία και Ολλανδία το θέμα είναι πολύ σημαντικό, το θέμα της επικουρικότητας. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ως πολιτική ομάδα για την για το νομικό εργαλείο, ο κανονισμός ε, εναρμονίζουν τις διαδικασίες. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και επομένως του αρέσει αυτό το νομικό μέσο, ο κανονισμός, η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς ε, τον εισηγητή που ήταν πολύ επικοδομητικός. Ε, είχαμε καλές συναντήσεις και πολύ σωστά είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των σημείων ε, μέσω των τροπολογιών του πρέπει να τύχουν ε, ευρεία υποστήριξη στην Επιτροπή. Ε, κάτι που δεν είναι προσωπικό. Ε, που θέλω να πω προ το συνάδελφο τη Επιτροπή των Περιφερειών. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με την Επιτροπή. Μπορεί να υποβάλει και κείμενα σε εμά. Αλλά πιστεύω ότι εδώ σε αυτό το χώρο, σε αυτή την Επιτροπή, είμαστε εκλεγμένοι και οποιοδήποτε είναι εκλεγμένος μπορεί να έρθει και να μιλήσει αυτήν την Επιτροπή. Ε, το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, είναι ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο. Συμφωνώ με τον εισηγητή για κάποια σημεία, αλλά όχι για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ, όταν κοιτάμε τις διεθνείς συμφωνίες, όταν κοιτάμε την ισορροπημένη προσέγγιση, τα πρότυπα CAPE, Αυτά είναι διεθνή πρότυπα. Και δεν είναι σωστό να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Γιατί είμαστε διεθνείς παίχτες, θέλουμε την ε, επιχειρηματικότητα, τον ανταγωνισμό, όλες οι επιχειρήσεις μας και οι απορικές εταιρείες προσπαθούν να ανταγωνιστούν. Ε, δεν θα πρέπει να αρχίσουμε τώρα να αλλάζουμε τους κανόνες. Επίσης συμφωνώ και για τα οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη. Ε, αναγνωρίζονται αυτά. Ξέρουμε πώς θα πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείε Για τα δεσιμπέλ, ε, η προηγούμενη συνάδελφο ε, είπε σωστά πράγματα. Μπορεί τελικά να έχουμε αεροσκάφη τα οποία μετά από 35 χρόνια ε, μετά από 35 χρόνια μάλλον πρέπει να κατέβουν ας πούμε τους αέρες. Το βασικό είναι τα περιφερειακά μας αεροδρόμια να αναπτύσσονται σωστά. Δεν θα έχουν πάντα τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη. Επίσης, δεν αναγνωρίζουμε το ρόλο των κρατών μελών. Θα πρέπει να πούμε και στα κράτη-μέλη ότι έχουν την ευθύνη για τις υποδομές και για το δυναμικό, γιατί, ας πούμε, ε, επιτρέπουν, ξέρω εγώ, γύρω από τα αεροδρόμια να φτιάχνονται κατοικίες, ε, θα πρέπει να τα δούμε και αυτά τα θέματα. Επίσης, όταν βλέπουμε τις νέες ε, τεχνικές στα αεροδρόμια, στους διαχειριστές ενέργειας κυκλοφορίας, ξέρετε ότι έχουν γίνει πολλές πρόοδοι τεχνολογικές, ε, προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια, μην το ξεχνάμε, και επίσης μπορούμε να καταλήξουμε σε καλά συμπεράσματα, όπως είπε ο συγητής, αλλά η Κομισιόν αλλάζει την οδηγία αυτή αφέρτα και την κάνει καονισμό. Ήταν οδηγία αρχικά. Και γιατί ήταν οδηγία. Γιατί υπάρχει το θέμα της επικουρικότητας, γιατί υπάρχουν τα θέματα τα τοπικά και δεν θέλω να περάσει σε καονισμό από την οδηγία χωρίς καμία συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να, παρα... να είναι οδηγία. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια θέματα με κάποια κρατημέλη, κάποιες ομάδες. Ορισμένοι θέλουν άλλα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε και ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Ε, με τις τοπικές συμφωνίες με τα, μεταξύ αεροδρομίων και ενδιαφερομένων ας πούμε, φορέων, τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Τέλος, ευχαριστώ τον εισηγητή για όλη την δουλειά του και γενικά νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Κυρία Ντεβεράκ. Για το θέμα του, νοή, του θορύβου, ε, συχνά μπορούμε να φτάσουμε σε δημαγωγικές δηλώσεις ε, και να φτάσουμε σε μία νομοθεσία άσχετη. Δεν συμφωνώ βέβαια με όλα τα θέματα του κυρίου Λάιχτφριντ. Ε, Παρ' όλα αυτά θέλω να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά που έκανε για αυτό το θέμα. Είπα και πριν ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω το άρθρο 10 για το δικαίωμα που προτείνει η Κομισιόν και τις διατάξεις που προτείνονται από το συνάδελφο στο σχέδιο έκθεσης. Ε, ε, μάλλον οι προτάσει του συναδέλφου είναι καλό συμβιβασμό. Ε, η εκτίμηση αυτών των μέτρων θα πρέπει να αφορούν τι τοπικέ αρχέ που γνωρίζουν πολύ καλά του τοπικού φορεί που δραστηριοποιούνται και δεν θέλουμε εδώ πέρα να αποφασίζουμε εδώ στην Επιτροπή στις Βρυξέλλες που είμαστε τόσο μακριά από όλα αυτά που συμβαίνουν στα τοπικά, στις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, συμφωνώ με, συναδέλφη με τους συναδέλφους για την προσφυγή στις ε, κατεξουδότηση πράξεις. Θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται ε, σε διαβούλευση με τους φορείς και τους εκπροσώπους τους. Οι εισαγωγές διατάξεων προσωρινών για τα μέτρα περιορισμού που έχουν υιοθετήθει σημαίνει ότι είμαστε στο ίδιο κύματος με τον εισηγητή. Για την ε, πρόταση του εισηγητή να μην πούμε βιαστικά σε ένα νέο ορισμό των αεροσκαφών που οριακά συμμορφώνονται, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την άποψή του. Τελευταίο σημείο. Εκεί που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον εισηγητή, με την ε, έννοια της υγείας των ε, περίοικων. Γιατί μπορούμε να βάλουμε ένα κριτήριο που δεν είναι ποσοτικό και είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η σχέση αιτία, αιτία, αιτίας αιτιατού ανάμεσα στο θόρυβο δηλαδή και στην υγεία των περίοικων. Μπορούμε να ανοίξουμε εδώ το κουτί της πανθόρας για αγωγές και τέτοια. Ε, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον σεβασμό τέτοιων κριτηρίων και δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες μελέτες είναι ισορροπημένες. Πέρα από το ερώτημα για το άρθρο 10, εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Πρώτον, ε, πέρα από την εξισορροπημένη προσέγγιση που τη γνωρίζω πολύ καλά, γιατί είχα συμμετάσχει και στις σχετικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της, ε, του Διεθνούς Οργανισμού ε, Πολιτικής Αεροπορίας. Ε, γνωρίζω λοιπόν και την απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, είναι σημαντικό να έχουμε κανονισμούς στο, ε, για το θόρυβο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ζήτημα της υγείας δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ή αόριστο. Είναι ένα ζήτημα κοινωνικό και επομένως τα, η προστασία των πολιτών από το θόρυβο είναι σημαντική. Τώρα, για την ισορροπημένη προσέγγιση. Πιστεύω ότι υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης εδώ. Γιατί τα μέτρα που λαμβάνουμε για την καταπολέμηση του θορύβου δεν επηρεάζουν ισότιμα όλους. Ε, ας σκεφτούμε για παράδειγμα το ζήτημα της ε, αρχής ο, ο Ριπένον πληρώνει κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και για το θόρυβο. Εκείνο ο οποίο προκαλεί το θόρυβο να είναι εκείνο ο οποίο θα πληρώσει. Όχι οι τοπικέ αρχέ οι οποίε έχουν ήδη μεγάλα προβλήματα με τον προπολογισμό του να πρέπει να αντιμετωπίσουν και αυτό το θέμα. Και το τρίτο ζήτημα, η πιστοποίηση για το θόρυβο των αεροσκαφών. Θεωρούμε πως δεν είναι καλό ε, μέτρο γιατί ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο θόρυβος κατά την πιστοποίηση των αεροσκαφών είναι πολύ διαφορετικός από τον θόρυβο ο οποίος προσλαμβάνεται από τους πολίτες όταν ένα αεροσκάφος ε, βρίσκεται στον αέρα. Επομένως θα είναι δύσκολο να... Ε, ε, ε μάλλον θα ε, υποστηρίξουμε συνολικά την έκθεση αλλά θα θέλουμε να ε, προτείνουμε τροπολογίες, γι' αυτό θα θέλαμε να καθυστερήσει η ε, προθεσμία μέχρι τις 28 ε, Σεπτεμβρίου αντί για τις 26. <laughs> Μιας και με ρωτάτε κατά πάση πιθανότητα η απάντηση είναι όχι, γιατί την είχαμε συμφωνήσει αυτή την ημερομηνία κατά τη συνάντηση των συντονιστών. Επομένως θα την διατηρήσουμε. 26 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Κρόσου. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θέλω να θυμίσω ότι μια που έχουμε διάφορε ημερομηνίε. Σε ό,τι αφορά γενικά το πακέτο, με μια άλλη έκθεση που δεν συζητάμε σήμερα, συνδέεται αυτό. Και να πω για τη συνάδελφό μας ότι χαίρομαι να ακούω την Επιτροπή Περιφερειών και την άποψή της για κάποια θέματα. Ναι, ακριβώς ε, είναι ένα θέμα ε, που χρειάζεται να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε διεθνώς ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις εθνικές αρχές αλλά και στις περιφερειακές. Και αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία της δουλειά μου. Γι' αυτό χαίρομαι. Ε, γι' αυτό που προτείνατε για το άρθρο 10 είναι σωστός δρόμος και επιδέχεται και κάποιες βελτιώσεις για να ενισχυθεί ακόμα ε, και σε σχέση με το αποτέλεσμα που υπάρχει σε διάφορες περιφέρειες να μην αλλάξουν οι κανόνες και να χρειαστεί από την αρχή να το ξανασυζητήσουμε. Γιατί αν έχουν βρει μια καλή λύση ε, οι περίοικοι, οι περιφερειακές αρχές και οι εθνικές αρχές και είναι ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε τα κριτήρια και να τα γκρεμίσουμε όλα. Ε, το θέμα της οικονομικής ε, αποτελεσματικότητας ή της γενικότερης, θέλω να πω, όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα θα πρέπει να έχουμε δύο πτυχές. Πρώτον, βέβαια το σύνολο του αεροσκάφου, το θόρυβο, τα θέματα υγείας, αλλά και πώς πολίτες αφορά. Γιατί άλλο είναι να έχεις δύο εκατομμύρια περίοικους και άλλο να έχεις δύο-τρεις χιλιάδες. Είναι πιο εύκολο ενώ να λυθεί το πρόβλημα και δεν θα πρέπει να το δούμε πάντα στην πηγή, αλλά ε, στην κατάληξη του, στον ίδιο τον πολίτη. Αυτά. Ε, πάντως γενικά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που ήδη έχουμε κάνει την προεργασία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ λοιπόν τον εισηγητή για τα οριακά συμμορφούμενα αεροσκάφη συμφωνώ πλήρω με την τροπολογία που προτείνεται, την 16. Αυτό είναι ο κατάλληλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. σω ορισμένοι από εμά θυμούνται το το θέμα του Haskit που είχε συζητηθεί πριν πολλά χρόνια, η διαφορά μεταξύ των ε, μηχανών της Rolls Royce ή της Pratt Whitney, τη θυμόμαστε πολύ καλά όταν προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας την προσέγγιση άλλων. Έτσι, η προσέγγιση που προτείνει ο θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη και με χαρά θα αναμείνω τις τροπολογίες που θα προταθούν. Η κυρία Μέη από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, το ζήτημα του θορύβου είναι ευαίσθητο και περίπλοκο το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε τοπικό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Ορισμένες αρχικές παρατηρήσεις για την έκθεση του κυρίου Λάιχτφριτ. Τέσσερις παρατηρήσεις. Το θέμα της υγείας και της ασφάλειας. Είναι αυτονόητο πως τα θέματα της υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο τοπικό επίπεδο, και η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει το θέμα των διαδικασιών που αγγίζουν τα, θέματα της υγείας και της ασφάλειας. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε την σχέση αυτής της οδηγίας με την οδηγία 2249 ε, για το περιβαλλοντικό θόρυβο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει πρόβλημα με τον όρο αποτελε... Ε, γενική αποτελεσματικότητα. Δεν είναι ξεκάθαρος αυτός ο όρος. Και όταν ε, υιοθετούνται κανόνες για τα οριακά συμμορφωμένα αεροσκάφη, πού θα θέσουμε το ε, όριο, πού θα πρέπει να επέμβουμε, θα είμαστε αυστηροί ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε ε, το όριο το, μάλλον λιγότερο από 10 δεσιμπέλ ε, θορύβου που γίνεται αντιληπτός. Εάν μειώσουμε κι άλλο αυτό το όριο, θα, δεν θα έχουν τη δυνατότητα οι τοπικές και οι εθνικές αρχές να παρεμβαίνουν. Τρίτον, και σημαντικό κατά την άποψή μου και για την Επιτροπή και για το Συμβούλιο είναι το ζήτημα του κατά πόσον θα έχει δικαίωμα η Επιτροπή να εξετάζει ε, τα θέματα αυτά. Όπως έχει ήδη υποθεί, η Επιτροπή δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τις τοπικές αρχές στη λήψη αποφάσεων. Χρειάζεται διαφάνεια και ε, αυτό μας οδήγησε να προτείνουμε το άρθρο 10 Και τελευταίο σημείο για το θέμα των της πράξεων. Είναι απαραίτητες για να επικυροποιούνται ορισμένες προβλέψεις της οδηγίες ε, της τεχνολογικής πρόοδου. Όπως αυτή κατοπτρίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές και από τα εγχειρίδια που εκδίδει η Διεθνής Οργάνωση πολιτική αεροπορία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να ε, κάνουμε ε, μέσω των κατεξουσιοδιώτης πράξεων πιο συμβατές τις προβλέψεις της οδηγίας. Αλλά χρειάζεται μια ε, σαφής διαδικασία έτσι ώστε να προσαρμόζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο με βάση αυτές τις προόδους και αλλαγές. Βρισκόμαστε στην διάθεση του εισηγητή και των μελών του Κοινοβουλίου για να συμφωνήσουμε τον καταλληλότερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, κύριο Λάιφ. Μάλλον πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λάιφ. Ε, πείτε μου αν μόνο εγώ το θυμάμαι αυτό, αλλά η Επιτροπή μου φαίνεται ότι πολύ επιλεκτικά επιλέγει αν θέλει να εφαρμόσει τους κανονισμούς του ΙΚΑΟ ή αν θέλει να μην τους εφαρμόσει κατά περίπτωση και τις, διεθνεί, και τις διεθνείς συμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Λάιφρυχ είναι ο ειδικός σας, μας τα πει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια που το αναφέρετε, εγώ δεν θα το έλεγα, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία της Επιτροπής είπε ουσιαστικά ότι ο λόγος για το άρθρο 10 ήταν λέει, για μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων των εθνικών αρχών. Αυτό το θεωρώ συμφωνία για τη συμβαστική μου πρόταση και αυτό αυξάνει ε, τη διαφάνεια. Οπότε δεν μιλάει πλέον για καταναγκαστικά μέτρα που δεν χρειάζονται από ό,τι φαίνεται. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ και χαίρομαι, έτσι το εκλαμβάνω. Ωραία, κατά τα άλλα δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά. Όπως είπα, όταν μου ανέλαβα αυτό το θέμα, είπα, Θεούλη μου, δεν πρόκειται να είναι απλό, αλλά δεν ήταν τόσο τραγικό όσο το φαντάστηκα. Γι' αυτό έχει να κάνει με την πάρα πολύ επικοδομητική στάση των συναδέλφων με τους οποίους έχω την ευκαιρία συνεργάζομαι και πραγματικά είχα και πάρα πολύ υψηλής ποιότητας δουλειά. Και αφού άρχισα στα αγγλικά θα ε, τελειώσω στα αγγλικά και νομίζω ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση η σιωπή είναι χρυσός. Λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου θυμίζω προθεσμία κατάθεση προ, ε, τροπολογιών, γιατί είναι πακέτο, γιατί ε, θα τη ψηφίσουμε στις 6 Νοεμβρίου εδώ το Δεκέμβριο νομίζω στην Ολομέλεια, αλλά θα εξαρτηθεί από διάφορες ε, ε, οροφές που πέφτουν, ε, ρογμές που ανακαλύπτουμε και άλλα τέτοια. τίνα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Θυμίζω ότι στις 3 η ώρα έχουμε μείνει ακρόαση για τις αστικές συγκοινωνίες, στις 3 ακριβώς, θα τα πούμε τότε. Και η κυρία την πρόεδρος του Κοινοβουλίου, θα ε, παρουσιάσει τους τέσσερις ομιλητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα λέμε το απόγευμα.